Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ θα ήθελα να αρχίσουμε πάρα αυτά και να ευχαριστήσω θερμά τους παρόντες και να σας πεθυμίσω ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται απευθεία στο τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου, όπως συνήθως. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο πρόεδρός μας, ο κύριος Σταυρακάκης, μας ζήτησε ένα δεκάλεπτο για να μας παρουσιάσει τη δική του γνωμοδότηση σήμερα για την ολοκληρωμένη πολιτική της θάλασσας, λίγο πριν το σεμινάριό μας, ενώ η ουσιαστική συζήτηση θα γίνει αύριο. Επίσης έχουμε και τους 28 δημάρχους από μικρά νησιά της Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό και τη γνωμοδότηση του κύριου Σταυρακάκη, στον οποίο θα δώσω πρώτα το λόγο για τη μικρή παρουσίαση αυτή, για να τιμήσουμε και τους προσκεκλημένους μας από την Ελλάδα. Αν συμφωνείτε με αυτή τη μικρή αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Uh, we have uh, Ως συνήθως ε, έχουμε διερμηνία από και προς 18 γλώσσες. Σημείο πρώτο της ημερήσιας διάταξης ε, διαθετήθηκε η έγκριση. Δεύτερο, οι ανακοινώσει της Προέδρου. Θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής μας να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία των δημάρχων που εκπροσωπούν τις μικρές ελληνικές νήσους. Επίσης να σας ενημερώσω ότι ετοιμάζουμε μία αντιπροσωπεία για τρεις γερμανικές πόλεις, Μανχάι, Πλουξεμπερκ και Χάιδελβέργη, 22 με 26 Ιουνίου, δηλαδή από αύριο ουσιαστικά μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος επισκέψεων που έχει εγκριθεί από το Προεδρείο μας και θα μεταβούν στην αντιπροσωπεία αυτή 8 συνάδελφοι, 3 Γερμανοί και στόχος όπως όλων των αποστολών των αντιπροσωπιών μας είναι να εξετάσουν διεξοδικά τις επενδύσεις των διαφορετικών ταμείων στο τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και ανταλλαγή απόψεων με τοπικούς φορείς για την πολιτική συνοχή και το μέλλον της. Ο Γιάνν Όλμπριχτ θα προεδρεύσει τις αντιπροσωπείες αυτής που θα μεταβεί στη Γερμανία. Και όπως ξέρετε σήμερα και αύριο έχουμε και την άτυπη υπουργική διάσκεψη στο Τολέδο, σήμερα για τη στέγαση. Κυρία Καλή Ντελή θα εκπροσωπήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αύριο θα γίνει η δεύτερη άτυπη υπουργική διάσκεψη για την ε, πολεοδομική ανάπτυξη, ανάπτυξη των πόλεων. Θα στείλουμε τριμελή αντιπροσωπεία, την κυρία Οκονή, τον κύριο Όλμπριχτ και την υποφερομένη. Πρώτο σημείο τη ημερήσια διάταξη, όπω είπαμε, θα είναι η παρουσίαση τη γραμματότητα του κυρίου Σταυρακάκη. Σα δίνουμε το λόγο, κύριε Σταυρακάκη. Πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους καλεσμένους μου, τους εκλεκτούς ε, δημάρχους των μικρών νησιών. Θα σας παρουσιάσω, είναι ιδιαίτερη μου τιμή και χαρά να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, αξιολόγησή της ως τώρα, προόδου και νέες, νέες προκλήσεις. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, η αηφόρος χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί ζωτική προϋπόθεση για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη όλης της Ευρώπης. Βασικοί τομείς όπως η αλία, η υδατοκαλλιέργεια και οι συνδεόμενες με αυτή βιομηχανίες, η ενέργεια, οι μεταφορές και ο τουρισμός αναπτύσσονται συνεχώς, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για τις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο, αυτοί οι τιμές αυξάνουν παράλληλα την πίεση για το θαλάσσιο περιβάλλον και το ζητούμενο είναι το πώς η ανάπτυξη αυτή θα είναι ισόρροπη προκειμένου να διασφαλίζει το επαγγελματικό μέλλον και τα εισοδήματα των πολιτών. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις απαντάει η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η οποία δεν παραλείπει να καλύψει τη σημαντική κοινωνική πτυχή της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής στις παράκτιες περιοχές, πτυχή η οποία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση της Ευρώπης 2020. Αυτό όμως που θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα είναι την καινοτόμο προσέγγιση που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία άλλαξε τον αποσπασματικό τρόπο διαμόρφωσης των πολιτικών και λήψης των αποφάσεων για το θαλάσσιο τομέα. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι όλα τα θέματα που συσχετίζονται με τους ωκεανούς και τις θάλασσες Ευρώπης διασυνδέονται και ότι όλες οι πολιτικές που συνδέονται με τη θάλασσα πρέπει να αναπτύσσονται συνεκτικά αν θέλουμε να αποκομίσουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και αυτή η προσέγγιση θα αναπτυσσόταν με πλήρη σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, εξού και ο πρώτος άξονας της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, που στοχεύει σε ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα μπορούν να αναλύσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φορέων και δράσεων προκειμένου να αναπτύξουν κοινά εργαλεία προς αξιοποίηση των συνεργειών και αποφυγή των συγκρούσεων. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν μέσα οριζόντιου σχεδιασμού, δηλαδή η θαλάσσια επιτήρηση, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η συνεκτική πηγή δεδομένων και πληροφοριών, τα οποία τέμουν τις τομεακές θαλάσσιες πολιτικές και στηρίζουν την αποκοινού χάραξη πολιτικής. Κάνοντας σήμερα ένα πρώτο απολογισμό για την υλοποίηση των στόχων, είναι αντιαφισβήτητο ότι η Όθουπου καλλιέργησε μια νέα κουλτούρα διακυβέρνησης, ενισχύοντας τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην υλοποίηση των δράσεων. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι περιφέρειες οι οποίες εσωμάτωσαν τις κύριες αρχές της, τα περιφερειακά τους προγράμματα, όπως η περιφέρεια της Δουνκέρνης ή η περιφέρεια της Βρετάνης, η οποία ανέπτυξε μάλιστα ειδικό πρόγραμμα για την παράκτια περιοχή. Στο σχέδιο γνωμοδότησης προσπάθησα να ενσωματώσω τα κύρια σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα αποτελέσουν τις κυριότερες προκλήσεις για το μέλλον της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής υπό το ειδικότερο πάντα πρίσμα της περιφερειακής πολιτικής και ανάπτυξης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στα εξή σημεία. Πρώτον, τη σημασία της αναγνώρισης της εδαφικής συνοχής από τη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ως νέα βάση για περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέσω της προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων καθώς και μέσω της βελτίωσης των συνδέσεων των απόκεντρων θαλάσσιων περιφερειών και των νησιών τόσο μεταξύ τους όσο και με την υπηρετική χώρα και με τα οικονομικά κέντρα. Στο ίδιο πλαίσιο θεωρώ ότι θα πρέπει να τονιστεί και η σημασία του μεταφορικού ισοδύναμου γιατί σε πολλές χώρες το κόστος των θαλάσσιων συγκοινωνιών ξεπερνά κατά πολύ αυτό των χερσαίων και πλήττει συνεπώ την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, την ανταγωνιστικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Μια τέτοια διάκριση αντίκειται σε οποιαδήποτε έννοια συνοχής, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφική. Δεύτερον, την ανάγκη ενίσχυση τη συνεργασία και της ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των θαλάσσιων περιφερειών ω μέσου για την αντιμετώπιση ορισμένων εκ των δυσκολιών που δημιουργούνται από την νησιωτικότητα. Τρίτον, την ανάγκη για διαμόρφωση τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών place-based local development strategies οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Τέταρτον, την ανάγκη για δημιουργία μιας υπηρεσίας εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οριζόντια διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τα νησιά προκειμένου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και οι ανάγκες τους να προωθηθούν και να λαμβάνουν υπόψη στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Και τέλος, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένες οι θαλάσσιες περιφέρειες, θα ήταν πιστεύω σημαντικό να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μέτρων για τη θαλάσσια ασφάλεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, αναμένω με ενδιαφέρον τις απόψεις σας σχόλια και παρατηρήσεις στη συζήτηση που θα γίνει αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Σας ευχαριστώ. Ωραία, ολοκληρώσαμε την παρουσίαση αυτή. Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο. Ευχαριστούμε κύριε Σταυρακάκη. Θα περάσουμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης το σεμινάριο για την απλούστευση της πολιτικής συνοχής. Θα θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι ότι είχαμε αποφασίσει το Μάρτιο να διοργανώσουμε αυτό το σεμινάριο στα πλαίσια της προετοιμασίας μας για τη λήψη αποφάσεων ως προς το μέλλον της πολιτικής συνοχής, καθώς και την εκπόνηση των κανονισμών για το μελλοντικό πλαίσιο αυτής της πολιτικής συνοχής. Επίσης είχαμε αποφασίσει να διοργανώσουμε το σεμινάριο και τη συζήτηση γιατί πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε σε διάφορες φάσεις της διαδικασίας απλοποίησης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της κρίσης. Οπότε είναι σημαντικό σημαντική αυτή η συζήτηση και ο απολογισμός των πρόσφατων πρωτοβουλειών της απλοποίησης. Για να δούμε ποιες από αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν, ποιες να μετριαστούν, ποιες έπεσαν στη λύθη μετά την πρώτη φάση της εμπειρίας μας. Βρισκόμαστε σε πλαίσια μιας ενδιάμεσης αναθεώρησης αυτής της απλούστευσης της συνοχής και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σημερινό σεμινάριο και η σχετική συζήτηση. Βέβαια, η βασική πρόκληση της απλούστευσης προέρχεται από την περιπλοκότητα της πολιτικής συνοχής και του πολυσύνθετου συστήματος διαχείρισης που τη χαρακτηρίζει. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι η πολιτική αυτή, η πολιτική συνοχής, ήταν ανέκαθεν πολύ φιλόδοξη. Ήθελε να εξυγχρονιστεί, να απλοποιηθεί και μάλιστα αυτή η φιλοδοξία τροφοδοτήθηκε από τον πολλαπλασιασμό των προκλήσεών της, από τη διεύρυνση που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διόγκωση της διοίκησης με αποτέλεσμα να αποδυναμωθεί η αποτελεσματικότητά της ε, ως προς την αντιμετώπιση τέτοιων διαδικασιών. Υπάρχει όμως και το θέμα της αποδοτικότητας και η ανάγκη της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας ε, που μας οθεί στην απλούστευση. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε και μια υγιή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Όλοι αυτοί οι λόγοι, λοιπόν, είναι πολύ εύλογοι. Δεν θέλουμε μία απλώς ε, μία πιο φιλική και αποδοτική πολιτική συνοχή, αλλά μία πολιτική συνοχή που θα ανταποκρίνεται σε όλα τα προαναφερθέντα κριτήρια. Θα πρέπει επίσης να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ διαφόρων στόχων και τομέων στους οποίους εφαρμόζεται, ελέγχεται και αξιολογείται η πολιτική συνοχή και επίσης θα πρέπει να βρούμε και την σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων φορέων και λειτουργίας του συστήματος. Για παράδειγμα, έχουμε τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όλα αυτά τα θεσμικά όργανα συνεργάζονται, αλλά α μην ξεχνούμε και τα άλλα επίπεδα που υπάρχουν, το εθνικό επίπεδο, το περιφερειακό, το τοπικό, που επίσης συνεργάζονται για την εφαρμογή για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Γι' αυτό η απλούστευση είναι πολύ δύσκολη, αλλά και απολύτως απαραίτητη. Και αυτό που τη δυσκολεύει είναι ότι θα πρέπει να υλοποιήσουμε τη φιλοδοξία και της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης και του Κοινοβουλίου, να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία της συνοχής. Γιατί θα μπορούσαμε να πλουσέψουμε τα πράγματα στέλνοντα απλώ τα κονδύλια στου εθνικού προπολογισμού. Αλλά πιστεύουμε ότι η κοινή διαχείριση έχει μεγάλη προσθεθέμενη αξία. Βέβαια, αυτή είναι και πιο περίπλοκη η κοινή διαχείριση από ότι η αποκεντρωμένη απλή διαχείριση. Επίσης, η απλούστευση αυτή θα, πρέπει να δημιουργήσει κινδύνους για τον κοινοτικό προπολογισμό, τον οποίο τροφοδοτούν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, όπω ξέρουμε. Δεν θέλουμε ταυτόχρονα να εγκαταλείψουμε το αντίθετο. Θα θέλουμε να τονώσουμε, να ενισχύσουμε μια καινοτόμα προσέγγιση της πολιτικής σε θέματα και financial engineering αλλά και επιλέξιμων προγραμμάτων. και να καταλήξουμε σε ένα αποτελεσματικό σύστημα και σχεδιασμού αλλά και εφαρμογής των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής. Η απλούστευση λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητη σήμερα θα πρέπει να λάβουμε καλύτερη υπόψη και τις διάφορες ιδιαιτερότητες ε, των ευρωπαϊκών περιφερειών, πόλεων και περιοχών και να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την πολιτική αυτή στα διάφορα επίπεδα και φάσεις της, ε, σεβόμενη ακριβώς ε, τη διαφορετικότητα και τις ιδιαιτερότητες των περιφερειών. Για τη συζήτηση αυτή έχουμε προσκαλέσει σήμερα δύο επιφανείς προσωπικότητες και έγκριτους εμπειρογνώμονες, τον καθηγητή Τζον Μπάκλεϊ από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, το Πανεπιστήμιο Στρασκλάιτ και τον Ρόλαντ Μπλομέιερ Δεν με ενημέρωσε όμως η γραμματεία ποιον εκπροσωπεί ο κύριος Ρόλαντ Μπλομέγερ. Χαίρομαι πολύ, μου λέτε το όνομα, αλλά δεν μου λέτε από πού έρχεται. Λέει Μπλομέγερ από τον Μπλομέγερ και Σάντσα, αλλά θα μας πει ο κύριος Μπλομέγερ τι ακριβώς ε, εκπροσωπεί. Ξέρουμε ότι σας ενδιαφέρει η πολιτική συνοχής και περιμένουμε τα φώτα σας. Έχουμε και τρεις ε, εκπροσώπους των εθνικών διοικήσεων, τον Μπράχαμ Watson από την Σκοτσέζικη κυβέρνηση που είναι επικεφαλής της ε, Αρχής Πιστοποίησης και της Χρηματοπιστωτικής Ομάδας ε, για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τον κύριο Μάρκ Καλούπα, που είναι Διευθυντής του Τμήματος ε, για το Συντονισμό της Εφαρμογής των Κοινοτικών Ταμείων στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολωνίας και έχουμε τον Γιάνν Γκρέγκορ, τον Διευθυντή του Τμήματος ε, Οικονομικής Διαχείρισης ε, του Αρμοδίου Υπουργείου της Τσεχίας. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Τζον Μπάχτλερ. Βέβαια, οι αρμόδιοι για το PowerPoint ε, βρίσκονται εκεί πίσω, οπότε καλύτερα να τους ενημερώνετε ότι θέλετε να περάσετε στην επόμενη διαφάνεια, γιατί δεν τους βλέπετε κατά πρόσωπο. Τζον, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το ενδιαφέρον εργαστήριο για την απλούστευση, απλοποίηση. Είμαι από το Κέντρο Ερευνών στο Πανεπιστήμιο Strathclyde στη Γλασκόβη που εξειδικεύεται σε έρευνα για τις περιφερειακές πολιτικές σε όλη την Ευρώπη. Στο σύντομο διάστημα που έχω στη διάθεσή μου θα θίξω αρκετά θέματα τα οποία αντιμετωπίζονται λεπτομερέστερα σε ένα συνοδευτικό έγγραφο παρουσίασης ε, που έχω. Θα καλύψω τρία θέματα κατά την παρουσίαση. Καταρχήν να δούμε τις τρέχουσες προσπάθειες απλοποίησης και να τις βάλουμε σε ένα πλαίσιο, βλέποντας τις ευρύτερες συζητήσεις για την απλοποίηση και επίσης θα πρέπει να δούμε τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν τα τελευταία χρόνια. Δεύτερον, θα ήθελα να κάνω μια αξιολόγηση αυτών των μέτρων απλούστευσης, θέτοντας κυρίως το ερώτημα ως προς τη χρησιμότητα. Πόσο πολύτιμα ήταν αυτά τα μέτρα που πρόσφατα εισήχθησαν με βάση ένα μείγμα πηγών πληροφοριών. Τέλος, θα ήθελα να κοιτάξουμε το μέλλον και τη συζήτηση που λαμβάνει χώρα για την πολιτική συνοχή μετά το 2013 που επικεντρώνεται εν μέρη στο θέμα της απλούστευσης κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο. Ας δούμε τα πρώτα θέματα. Στην πρώτη διαφάνεια παρακαλώ. Οι πρωτοβουλίες απλούστευσης μπαίνουν σε ένα πλαίσιο εδώ. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που συζητούμε όταν μιλάμε για απλούστευση στην πολιτική συνοχής αποτελεί μέρος ευρύτερη σειρά πρωτοβουλειών που ανελήφθησαν σε, πολλά, ε, ε, σε πολλούς τομείς της Κομισιόν για τη βελτίωση της διοίκησης την προηγούμενη δεκαετία. Υπάρχει αυτό το κυλιόμενο πρόγραμμα απλούστευση σε όλους τους τομείς πολιτικής για την κωδικοποίηση νομοθεσιών και υπάρχουν πολλές πράξεις και σελίδες που ελήφθησαν από τον κανονισμό τα τελευταία χρόνια. Έγιναν προσπάθειες για τη μείωση του διοικητικού κόστους σε σχέση με τη γραφειοκρατία, το red tape όπως λέμε στα αγγλικά γίνεται προσπάθεια αξιολόγησης του αντίκτυπου μεγάλων πολιτικών προτάσεων, θέτοντας την ερώτηση αν αυτές οι προτάσεις αποτελούν την καλύτερη επιλογή για την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου και υπάρχει και ολόκληρη σειρά άλλων πρωτοβουλειών όπως ε, εργασίες με τα κράτη-μέλη και διοργανικά μεταξύ των θεσμικών οργάνων για την καλύτερη ε, ρύθμιση. Στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε και αν δεν το θυμόμαστε να το θυμίσουμε ότι η Ατζέντα 2000 και οι σχετικές προτάσεις το τέλος της δεκαετίας του 90 επίσης έθεσαν τον στόχο της απλούστευσης της ε, διαχείρισης, της επίτευξης μεγαλύτερης ευελιξίας και της αποκέντρωσης της ε, υλοποίησης. Δεν είναι καινούργια πράγματα αυτά που συζητάμε τώρα δηλαδή και αν δούμε την Ατζέντα 2000 στο παρελθόν, ενώ βλέπουμε ότι έγιναν κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της απλούστευσης, η ε, εφαρμογή, βλέπουμε, η υλοποίηση έγινε πιο περίπλοκη. Υπάρχουν πιο αυστηρά κριτήρια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση των έργων κλπ. Γιατί Προσπαθούμε να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα στα πλαίσια των πολιτικών μας για να διασφαλίσουμε την έγκαιρη ε, χρηματοδότηση, την λογοδοσία στα οικονομικά θέματα και να καταλάβουμε καλύτερα τι επιδιώκουν τα προγράμματα στην πράξη. Και αυτό έχει να κάνει και με τις σημερινές μας συζητήσεις. Δηλαδή πώς ο στόχος της απλούστευσης ε, ως ένα βαθμό έρχεται σε σύγκρουση με άλλους στόχους που επίσης προσπαθούμε να επιτύχουμε στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Τώρα, αν μείνουμε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, βλέπουμε τις πρώτες εμπειρίες με την υλοποίηση 2000-2006. Τα κράτη-μέλη ασκούν πίεση στην ε, Κομισιόν για την απλούστευση της διαδικασίας εφαρμογής γιατί καταλάβαν αμέσω ότι νέες διαχειριστικές, διοικητικές προκλήσεις έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη και πολλές σοβαρές συζητήσεις οδήγησαν στην ανακοίνωση της Κομισιόν το 2003 για την, το συντονισμό, την ευέλικτη διαχείριση, απλούστευση και η προσπάθεια απλούστευση στον έλεγχο, στην υποβολή εκθέσεων, ε, στην ε, οικονομική διαχείριση. Όλες αυτές οι προτάσεις, ενώ εν μέρει επέτυχαν, νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι με μεικτά συναισθήματα αξιολογήθηκαν και έγιναν δεκτές από τα κράτη-μέλη. Εν μέρη λόγω του χρονοδιαγράμματος, γιατί το 2003 ήδη είχε λειτουργήσει η νέα προγραμματική περίοδος, είχε αρχίσει δηλαδή να εφαρμόζεται, οπότε ορισμένες αλλαγές δεν είχαν καλή σχέση κόστους ωφέλους. Στα πλαίσια του νέου πλαισίου διαπιστώθηκαν ότι υπήρχαν περιορισμοί στο τι θα μπορούσαν να επιτύχουν. Και ένα θέμα που διατρέχει όλη μου την ε, ομιλία είναι ότι κάθε μέτρο απλούστευσης έχει διαφορετική σημασία στα επιμέρους κράτη-μέλη διό, λόγω των διαφορών που υπάρχουν ε, σε θεσμικό πλαίσιο και στις διοικήσεις. Τώρα, ε, η αναθεώρηση, η μεταρρύθμιση της πολιτικής το 2006. Εδώ ενσωματώνουμε κάποια διδάγματα από την περίοδο 2000-2006. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε πολλά παρατήματα, υπάρχει πιο ευέλικτη προσέγγιση στην αξιολόγηση και η νέα αξιολόγηση της ε, συμμόρφωσης που στηρίζεται στην ε, ε, προσέγγιση με οικοδόμηση εμπιστοσύνη, όπως είδαμε στην προηγούμενη περίοδο. Και πάλι έγινε δεκτή με ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί αυξήθηκε ο φόρτος εργασίας στην προγραμματική, στα πλαίσια αυτής της περίοδου. Και πάμε έτσι στην επόμενη διαφάνεια. Τα πρόσφατα μέτρα απλούστευσης. Όπως και στην προηγούμενη περίοδο, η έναρξη των τωρινών προγραμμάτων συνέπεσε με ένα άλλο πακέτο απλούστευσης, αλλά σε αυτή την περίπτωση το έναυσμα για τα μέτρα αυτά είχε σχέση εν με την οικονομική κρίση και βλέπουμε μια ευρία αντίδραση της Κομισιόν με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για Ανάληψη Δράσης και το ε, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ε, Ανάκαμψης και ε, τις επενδύσεις που διοχετεύονται πια στην πραγματική οικονομία. Ο στόχος εδώ σε μεγάλο βαθμό ήταν η επιτάχυνση της ε, υλοποίησης με αυξημένη ευελιξία και απλούστευση των κανόνων. Και η Κομισιόν υπέβαλε σειρά συστάσεων που γρήγορα ακολουθήθηκαν από νομοθετικές τροπολογίες, ούτως ώστε να ε, καλυφθούν ε, νομοθετικά μέτρα, κανονισμοί και μη νομοθετικά μέτρα. Επόμενη διαφάνεια. Τώρα, στο συνοδευτικό έγγραφο, εμείς θέτουμε πάνω από 30 μέτρα νομοθετικού και μη νομοθετικού περιεχομένου και στην οθόνη έχω καταγράψει κάποιες βασικές κατηγορίες μέτρων απλούστευσης που εισήχθησαν μέσα μέσω αυτών των νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων. Για παράδειγμα, έχουμε αυξημένη ευελιξία ε, στο κλείσιμο των προγραμμάτων 2000-2006 σε ό,τι αφορά με ε, βελτίωση της ε, ημερομηνίας επιλεξιμότητας για τα μέτρα. Επίσης, ενθαρρύναμε επιτάχυνση των δαπανών σε περιπτώσεις όπου θα έπρεπε να υπάρχει ταχύτερη αντίδραση ε, λόγω της οικονομικής κρίσης. Επίσης ε, ε, το Jeremy, το Jessica, το τα μέτρα οικονομικής διαχείρισης financial engineering, βελτίωση επίσης των συστημάτων προχρηματοδότησης, ε, μεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες απλούστευσης ό,τι αφορά τους κανόνες επιλεξιμότητας, ευρύτερη χρήση ε, ποσών, εφάπαξ ποσών και απλουστευμένες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση, έλεγχο, ε, λιγότερες πληροφορίες ε, για μεγάλα προγράμματα που θα επαναλαμβανόταν κάθε φορά. Επίσης ε, για την αποδέσμευση των κονδυλίων, ευελιξία των, των τελικών ημερομηνιών και για την αποπληρωμή μεγάλων προγραμμάτων και έργων. Αυτό τι είναι μια πρώτη ανασκόπηση του πρώτου μέρους που θα ήθελα να δούμε και αφορά τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση της απλούστευσης όχι μόνο στην πρόσφατη περίοδο αλλά μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Επόμενη διαφάνεια. Στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης αυτό που θα ήθελα είναι να σας δώσω κάποιες πληροφορίες στο πόσο πολύτιμα ε, θεωρούνται αυτά τα μέτρα απλούστευσης δεν υπάρχει μία ε, άνωθεν συνεκτική ανάλυση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Οπότε ε, παίρνω διάφορες πηγές πληροφοριών για να καταλήξω σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Στη έκθεση στρατηγικής που υπευλήθη πέρσι, τα κράτη-μέλη εκλήθησαν να υποβάλουν έκθεση για τη χρήση που έκαναν των μέτρων, αλλά έχουμε εδώ μικτής ποιότητας πληροφοριών. Δηλαδή δεν είναι όλες οι πληροφορίες των κρατών μελών της ίδιας ποιότητας. Επίσης έγιναν κάποιες έρευνες και στηρίχθηκα σε αυτές για τις απόψεις των διαχειριστικών αρχών σε 16 κράτη-μέλη που υπάρχει από το πρόγραμμα IQNet, που είναι ένα δίκτυο για ανταλλαγή πληροφοριών, το οποίο διαχειρίζεται το δικό μου Ινστιτούτο, όπου οι διαχειριστές, οι μάνατζερ των προγραμμάτων εκλήθησαν να σχολιάσουν την αξία των επιμέρους μέτρων, την αποτελεσματικότητά τους και ε, σε διάφορα στάδια μέσα σε ένα χρόνο και εκλήθησαν να πούν τι πιστεύουν για τα μέτρα. Και για τους σκοπούς αυτού του εργαστηρίου κάναμε ένα ερωτηματολόγιο από τις διαχειριστικές Ρωτήσαμε τις διαχειριστικές αρχές δηλαδή με βάση ερωτηματολόγιο τι γνώμη είχαν για κάθε ένα από τα μέτρα. Και εκλήθησαν να τα ε, σχολιάσουν και να τα βαθμολογήσουν, δηλαδή υψηλής αξίας, μέτρια, χαμηλής. Το δίκτυο IQNet, το οποίο δεν φαίνεται πολύ καλά στη διαφάνεια, αλλά υπάρχει link ε, που παραπέμπει σε ιστοσελίδα στο κείμενό μου, ε, αναφέρει πολλές διαχειριστικές αρχές ε, εθνικού και περιφερειακού επίπεδου από τα 16 κράτη-μέλη. Τι λένε λοιπόν οι αρχές αυτές για τα πρόσφατα μέτρα απλούστευσης, πώς τα αξιολογούν. Εξετάσαμε πέντε ομάδες μέτρων, τα μη νομοθετικά, τροπολογίες στο γενικό κανονισμό, στο κανονισμό για τα κονδύλια, για τα ταμεία, τον εφαρμοστικό κανονισμό και τον προτινόμενο γενικό κανονισμό και τις τροπολογίες του. Το γενικότερο, το συνολικό μήνυμα που ελάβαμε είναι ότι εν πολύ τα μέτρα απλούστευσης ήταν αποτελεσματικά, εν μέρη τουλάχιστον. Ε, πολλές αρχές ε, τα χαιρέτησαν θερμά με θετική υποστήριξη, ε, ιδιαίτερα τις προσπάθειες να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση, να, αρθούν κάποια ε, εμπόδια και φραγμή στην υλοποίηση. Σε κάποιες χώρες και περιφέρειες βλέπουμε δε ότι υπήρξε μεγάλη συνεισφορά ε, για την καταπολέμηση της κρίσης από την πολιτική συνοχής μέσα από αυτά τα μέτρα. Επίσης, η πρόσληψη των μέτρων κυμαίνεται, διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, εξαρτάται από την κλίμακα των πόρων που διατίθενται, ε, την πολιτική ευρύτερων προσπαθειών που καταβάλουν τα κράτη-μέλη για την αντίδραση στην οικονομική κρίση. Η σημασία της πολιτικής συνοχής και των μέτρων αυτών εξαρτάται λοιπόν από ένα ευρύτερο μέτρο προσπαθειών που καταβάλουν τα κράτη-μέλη. Και Μάλιστα, ένας αριθμός αρχών εξέφρασαν ανησυχίες ε, πρώτον για τους κινδύνους ε, υλοποίησης λόγω των αυξημένων των πρόσθετων ευθυνών και η ε, περίπτωση να υπάρχουν προβλήματα στον έλεγχο μετά και ε, θεωρούν για την περίοδο αυτή ότι τα μέτρα έχουν καλές προθέσεις αλλά καμιά φορά ε, ξύνουν μόνο την επιφάνεια αυτού που χρειάζεται για την απλούστευση. Και πάλι αντανακλώντας εμπειρίες από το παρελθόν, το προχωρημένο στάδιο στην υλοποίηση κάποιων μέτρων θεωρούν ότι ε, δείχνει ότι ακόμα τα μέτρα δεν αξιοποιήθηκαν καλά γιατί η δυσκολία εισαγωγής τους ήταν μεγαλύτερη. Ε, επίσης, ο... το σύντομο χρονικό διάστημα ισχύω των μέτρων μπορεί να επηρεάζει αρνητικά ε, τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά τους ε, κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το υπόβαθρο αυτής της διαφάνειας υπάρχει και στο κείμενό μου, αλλά εδώ συνοψίζομαι ουσιαστικά τις αξιολογήσεις των μέτρων από τις διαχειριστικές αρχές. Οπότε ε, το μπλε τμήμα της διαφάνειας του γραφήματος ε, καλύπτει τα μέτρα τα οποία θεωρούν πολύτιμα οι διαχειριστικές αρχές. Αυτά που είναι με βυσινή, κοκκινοπό έχουν μέση αξία πάντα σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές και τα κίτρινα μέτρα είναι εκείνα των οποίων η αξία θεωρείται μάλλον χαμηλή από τις διαχειριστικές αρχές. Και αυτό που βλέπετε παντού είναι ότι ως επιτοπλίστων τα όλα τα πακέτα νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων θεωρούνται υψηλής ή μέσης αξίας σε διαφορετικό βαθμό από τις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών. Οπότε θετικά αποτιμώνται ε, εν μέρη τα περισσότερα μέτρα. Αν δούμε το κείμενο θα διαπιστώσουμε ότι κάθε ένα μέτρο ε, αποτιμάται διαφορετικά από τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τη σημασία του. Αυτά που αποτιμώνται καλύτερα αναφέρονται εδώ. Αυξημένη ευελιξία στο κλείσιμο ε, του, της περίοδου 2000-2006, προχρηματοδότηση το 2009, ε, απλουστευμένοι κανόνες ε, επιλεξιμότητας, ε, προϋποθέσεων, απλουστευμένη παρακολούθηση των ε, έργων και το, η δυνατότητα των κρατών μελών να μειώσουν τα ποσά που τα, τα διαχειρίστηκαν με παρατυπίες και που διορθώθηκαν σε επίπεδο κρατών μελών. Πάμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο μέρος της παρουσίασης. Αυτό που θα ήθελα τώρα είναι να μην μιλήσω για τις τρέχουσες ή πρόσφατες προσπάθειες απλούστευσης, και, αλλά να μιλήσω για το μέλλον. Όλες οι συνεισφορές στη συζήτηση, ε, στις στα ε, κείμενα των δύο επιτρόπων ε, για την περιφερειακή πολιτική πέρσι, στις άτυπες συνεδριάσεις των Υπουργών Περιφερειακής ε, Ανάπτυξης πρόσφατα στη Σαραγώσα και άλλες επίσης συνεισφορές στη μεταρρύθμιση της πολιτικής ε, ε, συνοχής. Όλοι λένε ότι θέλουμε απλούστερη και πιο αποτελεσματική πολιτική. Και ενώ υπάρχουν πολλές προκλήσεις που, στις οποίες εκεί που επικεντρώνονται αυτές οι συνεισφορές είναι να απλουστευτεί το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου διασφαλίζοντας την ε, κανονικότητα των πληρωμών. Προσπαθώντας να επιτύχουμε προόδου εδώ βλέπουμε διάφορες συζητήσει. τώρα να λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του ε, ε, χρηματοδοτικού κανονισμού και σε διάφορες ομάδες εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της Κομισιόν. Πολλά και διάφορα θέματα συζητώνται. Θα ήθελα όμως να επικεντρωθώ σε μια βασική πρόκληση που είναι η μεταρρύθμιση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου. Και βλέπουμε εδώ μια σειρά ιδεών που συζητώ, συζητούνται για να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Ένα ζήτημα είναι αν μπορούμε να έχουμε διαφορετικό σύστημα ελέγχου και διαχείρισης περνώντας από σύστημα τριών σε ένα σύστημα δύο επιπέδων με ενιαία αρχή πληρωμών και εκαθάρισης ελέγχου και κυλιόμενη διαδικασία εκαθάρισης και κλεισίματος των λογαριασμών. Ένα άλλο ερώτημα είναι αν μπορούμε να έχουμε διαφοροποίηση διαδικασιών, για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που κυμαίνονται ανάλογα με την κλίμακα της χρηματοδότησης, την εμπειρία των, των ε, υπεύθυνων για την ε, εφαρμογή, ε, τη διασφάλιση των διαδικασιών ή αν μπορούμε να έχουμε υψηλότερο ανεκτό επίπεδο σφάλματος. Το σχέδιο του οικονομισμού έχει μια διαφορετική πρόταση ανάλογα με τον τομέα της πολιτικής. Επίσης, εναρμόνιση των κανόνων επιλεξιμότητας με ενιαία σειρά κανόνων για όλα τα ταμεία και για όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι αν μπορούμε να προσαρμόσουμε τον κανόνα νησιν 2 για την αποδέσμευση που θα μπορούσε να χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο ή θα μπορούσε να είναι νησιν 3 ή θα μπορούσε να προσαρμόζεται σε ανάλογα με τις παρεμβάσεις. Ε, και τις ε, προϋποθέσεις και συνθήκες. Είναι πολλά βέβαια τα θέματα, πολύ περισσότερα από αυτά που σας είπα, αυτά που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Μέρος της συζήτηση για τις μεταρρύθμισεις αφορά τις αλλαγές στη διακυβέρνηση με ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο. Συζητούμε για την απόδοση, βελτίωση της απόδοσης με νέες προϋποθέσεις ε, υποβολής εκθέσεων, αξιολόγησης. Όλα αυτά βέβαια μπορεί να ε, δημιουργήσουν νέες πηγές περιπλοκότητας. Μπορεί να οδηγούν σε εξορθολογισμό και βελτίωση της απόδοσης, αλλά όλα αυτά δεν απλουστεύουν αναγκαστικά πάντοτε τις διαδικασίες. Επίσης, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω, μακριά από το μάντρα της απλούστευσης και να καταλάβουμε ότι το κόστος της διαχείρισης της πολιτικής θα πρέπει να εξεταστεί επίσης και να θέσουμε ερωτήματα. Μήπως είμαστε υπερβολικοί σε σχέση με την κλίμακα χρηματοδότησης. Κάποιες προτάσεις πρόσφατα λένε ότι σε σύγκριση με άλλες πηγές χρηματοδότησης από αναπτυξιακούς οργανισμούς ε, το διαχειριστικό κόστος της πολιτικής ε, συνοχής δεν διαφέρει πολύ. Ε, επίσης, αν μια πολιτική που συνεπάγεται επιμερισμένη διαχείριση, που αυτό αναγνωρίζεται το καλό, εάν εν είναι πιο σύνθετη. Τέλος, η ανάγκη να αναγνωρίσουμε τη, τη στάθμιση και να δούμε δηλαδή τα υπέρ και τα κατά, τη σχέση κόστους-οφέλους. Η αλλαγή αυτή καθ' αυτή συνεπάγεται κόστος πάντοτε, ιδιαίτερα σε χώρες και περιφέρειες όπου είναι μικρά τα ποσά της χρηματοδότησης, υπάρχει μια ανησυχία σε σχέση με τις επιπτώσεις μια ενδεχομένως ριζικής αλλαγής. Ιδιαίτερα αν οι ίδιες αρχές πρέπει να διαχειρίζονται δύο προγράμματα με διαφορετικά καθεστώτα διαχείρισης. Οπότε εδώ θα πρέπει να σταθμίσουμε τη σταθερότητα αφενός πιστεύω και την αποτελεσματικότητα από την άλλη. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπάχκλερ, για την πολύ πλήρη αξιολόγηση και παρουσίαση των προκλήσεων. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μπλομάιερ, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ, κύριε Ροντρίγκες, γιατί είσαστε μονίμως παρόν. Ε, δεν είναι συνηθισμένο να έρχονται οι, οι πρόεδροι στη συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναπτυξιακή, ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, αν θέλετε να πείτε κάτι ειδικά για τον νέο χρηματοδοτικό κανονισμό, α, έχετε το λόγο βεβαίως, μπορείτε να το κάνετε. Ε, και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ευχαριστώ, κυρία Χούπνερ. Μία σύντομη εισαγωγή να σας παρουσιαστώ. Ε, δουλεύω σε μια εταιρεία consultants που βρίσκεται στην ε, ισπανική περιοχή Καστίγια Λαμάντσα και ασχολούμε για την, ε, με τη διαχείριση ενός α, περιφερειακού προγράμματος. Ο κύριος Μπάχκλερ έθεσε το πλαίσιο. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας δώσω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία από συνεντεύξεις και από έρευνες που κάναμε τα τελευταία, τις τελευταίες δύο εβδομάδες Παρακαλώ, τη διαφάνεια. Η επόμενη διαφάνεια. Πολύ σύντομα, το περιεχόμενο της παρουσίασής μου. Θα παρουσιάσω τους στόχους, ε, τη μέθοδο που χρησιμοποίησαμε, την ανάλυση που κάναμε και κάποιες, ε, κάποια συμπεράσματα και συστάσεις τις οποίες προβήκαμε. πώς κατανοούμε το στόχο και τη συνεισφορά μας σε αυτό το εργαστήρι. Θεωρούμε ότι γίνεται μια επισκόπηση των μέτρων απλούστευσης που υιοθετήθηκαν ε, μέχρι στιγμής και αυτών που προτείνονται και που είναι ακόμα επιτάπητος προς συζήτηση ή που πρόσφατα συζητήθηκαν στο Κοινοβούλιο και με βάση τις συζητήσεις που κάναμε στην Ισπανία και κάποιες έρευνες που κάναμε να παρουσιάσουμε κάποιες εναλλακτικέ λύσεις για βελτίωση, τη διαχείριση και τον έλεγχο. Ε, ελέγχουμε, ε, εστιάζουμε στον έλεγχο και στην διαχείριση των ε, διαθωτικών ταμείων. Γιατί μας ενδιαφέρουν αυτά τα μέτρα απλούστευσης. Άρχισαμε να προβληματιζόμαστε από μία πρόσφατη έρευνα που παρήγγειλε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, ε, όπου ζητήσαμε από καμιά πενταριά ελεγκτικές αρχές που καλύπτουν ε, και τα 25 κράτη-μέλη, λέει ο μιλητής, για το πώς, ε, πώς αξιολογούν τα σημερινά διαχειριστικά και ελεγκτικά συστήματα. Στις γραφικές παραστάσεις της διαφάνειας βλέπετε ότι δύο τρίτα των ερωτηθέντων αισθάνονται ανήσυχοι με τις σημερινές ρυθμίσεις και θεωρούν ότι οι αποδέκτες μπορεί να αποθαρρύνονται από το σημερινό επίπεδο οικονομικού ελέγχου. Ε, ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι ένας από τους στόχους της πολιτικής συνοχής είναι να υποστηρίξουμε την καινοτομία. Και θα είναι και προτεραιότητα για το μέλλον. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες. Ε, ότι όσοι θέλουν να προωθήσουν την ε, καινοτομία απομακρύνονται από την ε, πολιτική συνοχή και ψάχνουν, ας πούμε, εθνικές ε, στηρίξεις και περιφερειακές στηρίξεις. Και οι διαχειριστές ασχολούνται περισσότερο με θέματα ελέγχου παρά με θέματα περιεχομένου τελικά. Αυτή ήταν έτσι η αίσθηση που προέκυψε από το, το 70% των ελεκτικών αρχών που έδωσαν τη γνώμη τους. Τώρα, γιατί θα σας μιλήσω. Κύριε Μπάχτλερ, ε, θέσατε το πλαίσιο, δεν θα πω τίποτα γι' αυτό. Θα μιλήσω για τις πέντε υιοθετήσεις μεταρρυθμίσεις, αλλαγές δηλαδή, και τις δύο που εκκρεμούν. Με βάση τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να διευκολυνθεί ε, η ροή της χρηματοδότησης στα πλαίσια της σημερινής ε, οικονομικής κρίσης και να είμαστε σίγουροι ότι τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής φτάνουν στους αποδέκτες, του δικαιούχους, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ε, πίσω από τις πολλές ε, αλλαγές που προτείνονται είναι να μειωθεί το γραφειοκρατικό άχθος, ε, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια με βάση τη σημερινή εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει και να μειώσουμε και κάποιε από τις απαιτήσει και προϋποθέσεις. Να κάνουμε τα πράγματα συνολικά δηλαδή πιο ε, απλά. Σύντομα, θα σας μιλήσω για τη μέθοδο. Πώς απαντήσαμε στις ερωτήσεις για το πόσο ε, αποτελεσματικά είναι τα μέτρα απλούστευσης μέχρι στιγμής. Καταρχάς, κάναμε μία έρευνα επιχάρτου, κοιτώντα όλες τις ε, τροπολογίες μία προς μία. Εν συνεχεία, κάναμε μία έρευνα τέλη του περασμένου μήνα και αρχές ε, του τωρινού μήνα, όπου 37 ελεκτικές αρχές από 19 κράτη-μέλη απάντησαν ε, και είπαν την άποψή τους για την αποτελεσματικότητα των προτινόμενων μέτρων ε, απλούστευσης. Γνωρίζω τη διαχείριση μόνο σε μία περιοχή. Προσπαθήσαμε λοιπόν να διαβρύνουμε λίγο το πλαίσιο και κάναμε και συνεντεύξεις με διαχειριστές των διαφορετικών ταμείων στην Ισπανία, στην Καστίγια Λεών, Αραγών και Καταλωνία και στην ε, Καστίγια Λαμάντσο, σε αυτές τις τέσσερις ε, ισπανικές περιοχές. Όσοι δεν γνωρίζετε αυτές τις ε, περιοχές, είναι τελείως διαφορετικές περιφέρειες. Είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη των προγραμμάτων. Τώρα για τα πορίσματά μας συνολικά. Καταρχάς βασιστήκαμε στην έρευνα που κάναμε επί χάρτου και επιβεβαιώθηκε όμως αυτό από τη συζήτηση που είχαμε με τους διαχειριστές. Συνολικά υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των ε, γενικών θα έλεγα τροπολογιών και των ειδικών τροπολογιών. Υπάρχουν και κάποιες ίσονος σημασία ε, ίσως σημασίας ε, τροπολογίες. Ε, έχουμε καμία εικοσαριά γενικές τροπολογίες που καλύπτουν όλους τους τομείς, ενώ οι ειδικέ τροπολογίες αφορούν συγκεκριμένα ταμεία εδαφική συνεργασία Φερρυπίν, ή μέσα για, τον, ε, για τους οικονομικούς κανόνες. Γιατί η διαφοροποίηση αυτή. Γιατί οι τροπολογίες που έχουν ειδική εφαρμογή έχουν λιγότερες επιπτώσεις για τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους, μια και αφορούν ένα συγκριτικά μικρότερο μερίδιο των κονδυλίων των ταμείων. Παραδείγματο χάρη πάρει τη Γερμανία τον Τζέρεμι, συγγνώμη, που είναι το λιγότερο από το 1% του συνολικού, α, των συνολικών κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής, η ενταφική συνεργασία 2,5%. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα ποσά είναι σχετικά περιορισμένα. Εν συνεχεία αναλύσαμε αυτές τις ε, τροπολογίες ε, σε σχέση με το στόχο τους για να βρούμε για ποιο λόγο προωθούνται αυτές οι τροπολογίες. Έχουμε καμιά 40, 39 πιο συγκεκριμένα ε, τροπολογίες. 21 αφορούν και εστιάζουν τη διευκρίνηση των ε, προϋποθέσεων που υπάρχουν σήμερα, να βελτιώσουν την κατανόηση, να καταλάβουν οι περιοχές των κρατών μελών περί πρόκειται. 13 αφορούν τη μείωση των ε, διοικητικών προϋποθέσεων και 17 αφορούν τις ε, οικονομικές ροές. Εξασφαλίζουν δηλαδή ότι τα κονδύλια με βάση τη σημερινή, το σημερινό πλαίσιο ας πούμε, οικονομικής κρίσης φτάνουν όντως στους πραγματικούς δικαιούχους και αποδέκτες. Τώρα, τι μας έδειξαν καταρχήν κάποιες έρευνες. Ζητήσαμε από τις ελεγκτικές αρχές να δώσουν αυτές ε, να δώσουν τις ε, απόψεις τους. Έγινε μια πρόσφατη ε, αξιολόγηση συμμόρφωσης, ε, όπου συμμετείχαν αυτές οι αρχές. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο θετικά. Θεωρούν ότι αυτά που, συγγνώμη, αυτά που υιοθετήθηκαν συνεισέφεραν στη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους Τα δύο τρίτα των άνθρωπων που απάντησαν θεωρούν ότι δεν υπάρχει αλλαγή στο διοικητικό άχθος. Ένα υψηλότερο ποσοστό, 20%, πιστεύουν ότι το διοικητικό άχθος έχει μάλιστα αυξηθεί. Μόνο το 17% θεωρούν ότι υπάρχει μείωση. Αυτά είναι για τις ε, τροπολογίες που έχουν ήδη υιοθετηθεί. Για αυτές που θα υιοθετηθούν φέτος τώρα, οι απόψεις είναι πολύ πιο θετικές. 60% πιστεύουν δεν θα υπάρξουν αλλαγές, αλλά το 1 τρίτο παρόλα αυτά πιστεύει ότι πράγματι αυτές οι αλλαγές θα μειώσουν το γραφειοκρατικό άχθος. Καλύτερη δηλαδή αποτίμηση. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ένα άλλο ερώτημα που θέσαμε στο πλαίσιο της έρευνας είναι ο δεύτερος βασικός ε, λόγος. Φτάνουν τα λεφτά στους δικαιούχους με πιο αποτελεσματικό τρόπο, γρηγορότερα ας πούμε, ε, με πιο ευρύ, υπάρχει μια πιο ευρύ κάλυψη, υπάρχουν περισσότερα θέματα που καλύπτονται. Και πάλι οι απαντήσεις δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές. 72% των ερωτηθέντων, των ελεκτικών αρχών δηλαδή που απάντησαν, θεωρούν ότι δεν υπάρχει αλλαγή σε σχέση με τα κονδύλια που φτάνουν στους δικαιούχους, με μια επιφύλαξη ότι κάποια από τα μέτρα όμως είναι αρκετά πρόσφατα και Πρέπει λοιπόν να τους αφήσουμε λίγο χρόνο για να επηρεάσουν την κατάσταση. Αλλά αυτό απεικονίζει σε κάποιο βαθμό τις προσδοκίες των ελεκτικών αρχών. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Να πω δύο λόγια για τις συναντεύξεις μας στις τέσσερις διαφορετικές ισπανικές ε, περιφέρειες. Συνολικά υπήρχαν αρκετές επικρίσεις, όπως σας είπα, για αυτά τα μέτρα που υιοθετήθηκαν μέχρι σήμερα και για αυτά που συζητώνται με σκοπό να υιοθετηθούν ε, και που πιστεύουν ότι γενικά το γραφειοκρατικό άχθος δεν έχει ουσιαστικά μειωθεί. Ένα από τα προβλήματα που προέκυψε από τη συζήτηση με τις ε, περιφέρειες είναι το θέμα της επανάληψης των ελέγχων Πολλές αρχές μίλησαν για αυτό το πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα που συζητήσαμε διαμακρών αφορά την πρόσφατη αξιολόγηση συμμόρφωσης για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα. Εδώ υπήρχε μια θετική προσδοκία και πολλοί διαχειριστές θεωρούν ότι αυτή η αξιολόγηση είναι καλή. Ε, γιατί τώρα οι κανόνες είναι πολύ πιο ξεκάθαροι και δεν θα εκπλαγούν από αλλαγή των κανόνων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Από τους πρώτους ελέγχου, η εμπειρία είναι ότι αυτή, αυτή η αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν αύξησε παρόλα αυτά κατά ανάγκη την εμπιστοσύνη και επομένως κάτι υπάρχει εδώ που λείπει. Ένας, υπάρχει ένας ε, λοιπόν κρίκος. Ε, το, συζητήσαμε το θέμα της αναλογικότητας. Ε, κάποιες από τις ε, περιοχές που επισκεφτήκαμε, όπως η Αραγώνα, έχουν μικρότερα προγράμματα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ισπανικές περιοχές με μικρά προγράμματα. Και εκεί δεν αισθάνονται οι αρχές ότι οι προϋποθέσεις που τους αφορούν είναι διαφορετικές από τις περιοχές που, που τρέχουν μεγαλύτερα προγράμματα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Ένα από τα θέματα που μας υποδείχτηκε είναι ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να υπάρχουν αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί ελέγχου σε κάθε το επίπεδο. Πολλές ε, περιοχές, περιφέρειες μας είπαν ότι τα, τα ίδια θέματα αξιολογούνται από τους ελέγχους ας πούμε των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αρχών και τα ίδια ακριβώ πράγματα ελέγχει πάλι και η Επιτροπή με το ελεγκτικό συνέδριο. Ίσως θα μπορούσαμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα αν υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός. Βέβαια υπάρχει και ένα θέμα με την ερμηνεία των ε, κανόνων του, του κανονισμού σε εθνικό επίπεδο. Πάμε στο οριζόντιο επίπεδο. Οι αρχές των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων. Ο γενικός ε, κανονισμός διαφοροποιεί ξεκάθαρα τα καθήκοντα των τριών αρχών. Αλλά στις ε, περιφέρειες υπάρχει αίσθηση ότι δημιουργούνται επικαλύψεις μεταξύ των ελέγχων που γίνονται σε διάφορα επίπεδα. Από μια έρευνα που κάναμε πρόσφατα, που την παρήγγειλε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, βρήκαμε ότι τα κράτη-μέλη εδώ εμπλέκονται. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διευκρινίσουν ε, στα πλαίσια της δικής τους διοίκησης ε, πώς θα αποφευθούν αυτές οι επικαλύψεις. Σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται περισσότερα από ένα κράτη-μέλη, παραδείγματος χάρη διαχειριζόμαστε Έχουμε μάλλον ε, μία... Έχουμε ένα πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας. Έχουμε, μπορεί να έχουμε μία αρχή ας πούμε, διαχειριστική που βρίσκεται στο ένα κρατός μέλος, ενώ μία αρχή πιστοποίηση σε ένα άλλο κρατό μέλο. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα συντονισμού. Οι προτάσεις ε, της Κομισιόν για αλλαγές μας εξέπληξαν και το, υπόδει, το υπέδειξε αυτό το σημείο και το Κοινοβούλιο ότι δεν υπάρχει αρκετή διαβούλευση για κάποιες από τις τροπολογίες. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι δεν έγινε αξιολόγηση ε, για τα ρυθμιστικά μέτρα, δεν υπάρχει εξωτερική πραγματογνωμοσύνη και περιορισμένος γενικά περισμένες διαβουλεύσεις. Μία από τις προτάσεις της Κομισιόν το λέει κιόλα ότι λόγω του κατεπήγοντος χαρακτήρα δεν υπήρξε καθόλου α, διαβούλευση για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Θέσαμε αυτό το ερώτημα και στις ε, ελεκτικές αρχές, πέρα από τις ε, έρευνες όπου το θέσαμε και ε, πάνω από το 50% μας είπαν ότι ναι, έχουν δώσει τη γνώμη τους, το 1 τέταρτο περίπου, όχι το 1 τρίτο. Θεωρούν ότι έδωσαν τη γνώμη του και ότι η γνώμη τους έχει ληφθεί υπόψη. Στη δική μου περιφέρεια, κάτι που βρίσκω παράδοξο είναι ότι η πρόσφατη άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Περιφερειακής Πολιτικής δεν ε, βασίστηκε στις συζητήσεις που έχουν γίνει στις περιφέρειες. Τουλάχιστον στη δική μου περιφέρεια υπήρχαν κάποιες απόψεις που δεν ελήφθησαν υπόψη. Ίσως σε εθνικό επίπεδο αυτή υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση. Αλλά καλό θα ήταν στις επόμενες συνεδριάσεις να υπάρχει μια καλύτερη ε, διαδικασία διαβούλευσης όπου η άμεση ε, εμπειρία των ανθρώπων που εφαρμόζουν ε, τα προγράμματα και παίρνουν τα κονδύλια για την εφαρμή των προγραμμάτων λαμβάνεται υπόψη. Συμπεράσματα γενικά. Η εμπειρία, η, μας είναι ότι οι τροπολογίες ε, είναι λίγο σημαντικές για τις αρχές, για τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους. Και ο καθηγητής ανέφερε προηγουμένως ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Αυτό προκύπτει από τις διαβουλεύσεις μας. Στις μελλοντικέ τροπολογίες, ας λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν, υπάρχουν ε, έτσι, μειονεκτήματα ε, και θα θέλαμε να διορθωθούν στην περίοδο προγραμματισμού. Υπάρχει περιθώριο για τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους με τη μείωση των προϋποθέσεων και με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνόταν η διοχέτευση των ε, κονδυλίων των διαχωτικών ταμείων. Οι διαχειριστές ε, των προγραμμάτων ασχολούνται περισσότερο με τον έλεγχο. Παραδείγματος χάρη όταν ας πούμε, προετοιμάζονται πολύ τα προγράμματα, ε, φερρυπίν, όταν υπάρχουν προγράμματα καινοτομία, θα έπρεπε να δίδονται κατάλληλοι πόροι για να προετοιμάζονται καλύτερα αυτά τα προγράμματα και να μην ασχολούνται μόνο με τον έλεγχο οι διαχειριστέ. Συστάσει. Συμφωνώ με τον καθηγητή Μπάχτλερ. Αναλογικότητα. Να διερευνήσουμε τις ευκαιρίε για να ενδυναμώσουμε την σχέση της αρχής ε, αναλογικότητας και της ενσωμάτωσής της στον ε, γενικό κανονισμό. το θέμα της ε, εμπιστοσύνη. Να δούμε διαφορετικά τα μικρά προγράμματα από τα μεγάλα. Στα μικρά προγράμματα προωθούνται εξαιρέσεις. Παράδειγμα, είναι κάτω από τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. συγγνώμη, 750. Για τον έλεγχο. Υπάρχουν, υπάρχουν τα δύο επίπεδα ελέγχου, το οριζόντιο και το κάθετο. Σε οριζόντιο θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των τριών αρχών, ούτω ώστε να μην έχουμε επικαλύψεις με των τριών επιπέδων, μεταξύ των τριών αρχών δηλαδή των διαφορετικών ταμείων. και να δούμε πώς κάποιες προϋποθέσεις αρχίζουν να ισχύουν μόνο όταν προκύψει το πρόβλημα. Και να μην τα ελέγχουμε κάθε χρόνο για τα διαφορετικά ταμεία. Στο κάθε το επίπεδο τώρα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων ε, που διεργούν το έλεγχο, τον έλεγχο. Η συνθήκη μας δίνει τις δυνατότητε να κάνουμε κοινού ελέγχου μεταξύ του ελεγκτικού συνεδρίου και των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Προ το παρόν δεν συμβαίνει καθόλου. Υπάρχει τώρα μια πιλωτική προσπάθεια ευπρόσδεκτη, όπου η Ολλανδία, η Τσεχία και η Δανία κάνουν μια τέτοια προσπάθεια. Θα έπρεπε όμως να εντατικοποιήσουμε αυτή την προσέγγιση, ούτως ώστε να μεγιστοποιήσουμε τον συντονισμό στους ελέγχους. Τέλος. Πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Πώς θα βελτιώσουμε περαιτέρω, πώς θα τροποποιήσουμε περαιτέρω το πλαίσιο στο μέλλον. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερο αξιολογήσεις ρυθμιστικού χαρακτήρα ρυθμιστικών επιπτώσεων και να εμπλέξουμε περισσότερα κράτη-μέλη. Το μέλλον της ε, πολιτικής συνοχής ε, βασίζεται σε ένα ισχυρότερο διάλογο. Το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βότσον, θέλετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Um, ευχαριστώ. Είμαι επικεφαλής της αρχής πιστοποίησης και οικονομικής ομάδας τη Σκοτσέζικη κυβέρνησης. αλλά δεν εκπροσωπώ εδώ τη Σκοτσέζικη Κυβέρνηση. Αλλά θα ήθελα να σα μεταφέρω την πρακτική μου πείρα και την ε, εμπειρία που είχα και με άλλες ε, αρχές πιστοποίησης σε διάφορες χώρες. Είμαι ελεγκτής, ε, εργάζομαι για την σκοτσέζικη κυβέρνηση και ασχολούμαι και με το λογιστικό έλεγχο, οπότε αισθάνομαι μεγάλη συμπάθεια και συμπαράσταση για τις αρμόδιες αρχές που παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα. Φυσικά υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα από τις νέες προτάσεις. Το πρώτο που θα έλεγα είναι ότι δεν μπορεί κανείς να τους ευχαριστεί όλους πάντοτε, αλλά ας προσπαθήσουμε να ικανοποιούμε τους περισσότερους ως επιτοπλίστων πακέτο απλούστευσης ήταν περιορισμένης χρήσης για μας. Περιορισμένης με την έννοια ότι δεν εξυγχρόνισε καθόλου την διαχείριση των προγραμμάτων. Μας δυσκόλεψε μάλλον. Βέβαια μας έδωσε τη δυνατότητα να καναλιζάρουμε κονδυλία σε συγκεκριμένους τομείς. Μπορέσαμε ας πούμε να κατευθύνουμε χρήματα σε ε, οικονομικά από ενεργειακή άποψη σπίτια και αυτό ήταν σημαντικό. Είχαμε τον Τζέσικα, Τζέρεμι κλπ. Είχαμε τη δυνατότητα να παραδώσουμε ένα πρόγραμμα Αλλάζοντά το στα μισά. Αυτό είναι και περίπλοκο και δύσκολο εγχείρημα ιδιαίτερα όταν ε, αποδεσμεύομαι μεγάλα κονδύλια στην αρχή δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε διακρίσεις μεταξύ ε, αυτών που υπέβαλαν αίτηση πριν ή αργότερα. Οι αλλαγές λοιπόν είναι ε, ευπρόσδεκτες, ε, αλλά δυσχεραίνεται η δυνατότητα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας. Εγώ συμφωνώ με την απλούστευση της διαχειριστικής αρχής των αρχών ελέγχου, αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνουμε σε περιφερειακό επίπεδο στα κράτη-μέλη και είμαι επιφορτισμένος με το σύστημα ελέγχου. Βεβαιώνομαι ότι όλες οι αρχές και τα επίπεδα ελέγχου δεν ελέγχουν το ίδιο πράγμα για να αποφεύγουμε επικαλύψεις. Δεν θέλουμε η αρχή πιστοποίησης να καλύπτει όλη την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου, όλες τις περιφέρειες, υπάρχουν συγκεκριμένα επιμερισμένα καθήκοντα και λειτουργούν καλά. Η αλλαγή ενός τέτοιου συστήματος που έχει ρονταριστεί αποτελεί ριζοσπαστική αλλαγή. Και μπορούμε μέχρι το 2013 τα αφήσουμε όμως έχει και να κάνουμε τροποποίησεις μετά. Βέβαια μετά θα, κάποια στιγμή θα... Ε, ε, ε, θα ήταν ε, καταστροφικό να έχουμε συστήματα που να λειτουργούν ταυτόχρονα. Το ένα να τελειώνει και το άλλο να αρχίζει. Ε, Επίση θα πρέπει να έχουμε απλούστευση στη διαδικασία παράτασης των προγραμμάτων, να έχουμε μια δυνατότητα να κλείσουμε όπως πρέπει τα προγράμματα. Δεν, θα, δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε δύο τελείως διαφορετικά συστήματα που να τρέχουν ταυτόχρονα, γιατί αυτό είναι περίπλοκο, δαπανηρό και βέβαια οι ίδιοι θα είναι που θα ε, δραστηριοποιούνται και στα δύο επίπεδα και στα δύο προγράμματα. Δεν θα έχουμε δύο χωριστές ομάδες. Ο τύπος στο Ηνωμένο Βασίλειο... Ε, βρήθη περικοπών του προϋπολογισμού, από περικοπές του προϋπολογισμού για του χρόνου και τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι ότι η Κομισιόν θα πρέπει να θέσει λοιπόν ένα δύσκολο ε, ερώτημα στον εαυτό της. Χρειάζονται τόση πολύ έλεγχοι και παρακολούθηση, να υπάρχουν δύο-τρεις γενικές διευθύνσεις που να το κάνουν αυτό. Πρέπει να το σκεφτούν πολύ. Ε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και το λογιστικό έλεγχο, ε, πριν από δύο εβδομάδες είχαμε ε, πέντε συνολικά ελέγχους, λογιστικούς και μη, σε μια οργάνωση 50 ανθρώπων ε, και έμειναν όλη τη μέρα. Δεν ε, είναι καλό αυτό το μήνυμα. Αυτό δείχνει ότι δεν γίνεται ομαλά η διαχείριση και ο έλεγχος και ότι διασπαθίζονται πόροι. Η απλούστευση είναι συνεχής διαδικασία. Από τότε που άρχισαν τα προγράμματα μας απασχολεί. Οι αλλαγές χάρη των αλλαγών δεν εξυπηρετούν δεν έχει κανένα νόημα να ξαναγυρίσουμε σε παλιά συστήματα. Θα πρέπει να κάνουμε αλλαγές ριζοσπαστικές, να μην γυρίσουμε στην περίοδο 2000-2006. Είναι παράλογο. Ένα από τα μεγάλα θέματα που μας επηρεάζουν είναι η διαχείριση του κινδύνου. Η ανάθεση του ελέγχου στα κράτη-μέλη είναι καλό πράγμα στο βαθμό που γίνεται καλά η διαχείριση, ε, στο βαθμό που ο λογιστικός έλεγχος γίνεται ε, σωστά ε, και όχι στο τέλος της εξαετούς περίοδου να μας πούν δεν συμφωνούμε με αυτά που κάνατε. Όλα τα κράτη-μέλη, η αγγλική, η ουαλική κυβέρνηση, η σκοτική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντήσουν στο τέλος το ερώτημα σχετικά με τα έργα, εάν αυτά είχαν νόημα, εάν ήταν αποτελεσματικά. Ε, επίσης, όταν πρόκειται για μεγάλα έργα, ε, θα πρέπει να αναλάβουμε και έναν κίνδυνο. Μπορεί να κάνουμε κάποια δουλειά και μετά να απορριφθούν από την ε, Κομισιόν. Είναι ένας κίνδυνος αυτό, ένα ρίσκο. Υπάρχουν πλεονεκτήματα, υπάρχουν ε, και μειονεκτήματα στην απλούστευση. Κάθε περιφέρεια τα χρησιμοποιεί κάπως διαφοροποιημένα τα καινούργια ε, συστήματα. Δεν μπορούμε να ικανοποιούμε τους πάντες πάντοτε, όπως σας είπα, αλλά Ε, υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολα και λεπτά θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή η διάκριση ας πούμε, μεταξύ κάποιας παρατυπίας και της απάτης ε, ως επιτοπλίστων πρόκειται για παρατυπίες. 99% των περιπτώσεων βλέπουμε ότι δεν έχουμε απάτη. Όμως ο τύπος ε, αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά τα θέματα αυτά και μιλά πάντοτε για απάτη. Θα είναι λίγες οι περιπτώσεις απάτης. Θα πρέπει ίσως να βρούμε μια διαφορετική λέξη, ε, όχι παρατυπία. Ναι στην απλούστευση λοιπόν, αλλά νομίζω ότι δεν είναι σωστό να κάνουμε ριζικές και ευνίδιες αλλαγές σε μια νυχτή, αλλά σταδιακά βήματα. Χρειάζεται χρόνος για την εφαρμογή των νέων πραγμάτων, των νέων συστημάτων. Δεν μπορούμε δηλαδή στα μισά ενός προγράμματος που τρέχει να πούμε θέλουμε να τα αλλάξουμε, να κάνουμε κάτι άλλο. Θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε τον επόμενο χρόνο, να, έχουμε, να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να ε, εφαρμόσουμε και να ε, συστήσουμε τις νέες διαδικασίες και συστήματα. Αυτά είχα να σας πω, ελπίζω να είχαν κάποια ωφέλεια για σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάρε Καλούπα από την Πολωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εκφράσω την άποψή μου. Η πολιτική συνοχής δεν είναι ένας ε, ιδανικός μηχανισμός. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, μίλησαν για τις δυσκολίες ε, με τα, με συστήματα ελέγχου και τα συστήματα διαχείρισης. Θα μιλήσω και εγώ για αυτά τα συστήματα. Η πολιτική συνοχής έχει την ατυχία να βρίσκεται στο σταυροδρόμι διαφόρων και πολυπίκυλων ευρωπαϊκών ε, πολιτικών. Οι διάφορες ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες προσπαθούν να ακολουθήσουν τις διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας υψηλός κίνδυνος σφάλματος. Λόγω της φύσης της πολιτικής συνοχής και του μεγέθους της. Η πολιτική συνοχής είναι ένα τομέα όπου οι στόχοι άλλων πολιτικών α, ε, επηρεάζουν και υπάρχει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό σφάλματος. Γίνεται μια συζήτηση για την αύξηση του αποδεκτού ποσοστού σφάλματος πάνω από το 2%. Όμως αυτό θα σήμαινε ότι αντιμετωπίζουμε την αρρώστια ε, αντιμετωπίζοντας τα συμπτώματα και όχι τις αιτίες της αρρώστιας. Και γίνεται μια προσπάθεια απλοποίησης της πολιτικής συνοχής. Μερικές από αυτές τις αλλαγές ε, τις καλωσορίζουμε. Για παράδειγμα, δια, παράταση της ε, περίοδου για την εφαρμογή της προηγούμενης πολιτικής. Επίσης, τη δυνατότητα δυνατότητας υποβολής των αιτήσεων προκαταβολής. Αυτά τα στοιχεία μας αρέσουν. Βέβαια θα πρέπει να, διαπιστώσουμε ότι μέχρι στιγμής προσπάθειες απλοποίησης της πολιτικής συνοχής μας υπενθύμησαν κάποιες προσπάθειες <laughs> να ε, θεραπεύσουμε τη φυματίωση με καλύτερη υγιεινή του στόματος. Για παράδειγμα, πλένοντας καλύτερα τα δόντια μα. Φυσικά η υγιεινή του στόματος είναι πολύ σημαντική, αλλά σίγουρα δεν εξυπηρετεί τη θεραπεία της φυματίωση, Κάπως έτσι μας φαίνονται μερικές προσπάθειες απλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Δεν είναι όλες οι προσπάθειες αυτές της απλοποίησης αποτελεσματικές. Θα πρέπει να δούμε Ποιε διορθώσει θα πρέπει να γίνουν, πού θα πρέπει να βελτιωθεί ο έλεγχος και το φάσμα των δυνατοτήτων αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικά μεγάλο δυστυχώς και πολλές φορές τα κράτη-μέλη αδυνατούν να αποφύγουν τέτοια λάθη σε ό,τι αφορά τις διορθώσεις και τα λογιστικά τους. Επίσης, αντί να αυξήσουμε την ανοχή του σφάλματος, να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα σφάλματα που υπόκεινται σε χρηματικές και οικονομικές κυρώσεις. Θα πρέπει να καθορίσουμε λοιπόν το εύρος τους, αντί να αυξήσουμε το περιθώριο ανοχής. Το τελευταίο σχέδιο κανονισμού, του χρηματοπιστωτικού κανονισμού μας δημιούργησε αρκετές ανησυχίες. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας θορύβησε κάπως. Γιατί φαίνεται να προεξοφλεί ορισμένες διαρθρώσεις σε ό,τι αφορά τον έλεγχο με την ε, εισαγωγή αυτού του συστήματος του Annual Clearance of Accounts, της ετήσιας καθάριση των λογαριασμών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς, ε, η πρόφαση για την πρόταση του κανονισμού είναι η απλούστευση. Κατά τη γνώμη μας όμως, το σύστημα αυτό δεν βαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση, δεν βαίνει προ την κατεύθυνση τη απλούστευση. παρόλο που αυτό ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμ, επιτυχαίνει κάποια εναρμόνιση για κάποια απλούστευση ό,τι αφορά το συμψηφισμό και την εκαθάριση των λογαριασμών, ιδιαίτερα στην κυνηγιορική πολιτική. Αλλά αυτό το σύστημα δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στου ελεκτικού μηχανισμού των κρατών μελών. Ενώ αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να βελτιώσουμε στα κράτη-μέλη, την ακρίβεια αυτών των ελέγχων. Με την πρόταση αυτή του κανονισμού του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αυξηθούν τα σφάλματα αντί να μειωθούν και να βελτιωθεί η χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια πρόταση δεν είναι απλούστευση, απλώς στέλνει το μπαλάκι στις ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών και στις διαχειριστικές αρχές και μάλιστα αυξάνει την πίεση προς τις ε, αρχές αυτές για να ελέγξουν καλύτερα τις δαπάνες τους. Οπότε θα πρέπει να διαρωτηθούμε τι θα πρέπει να ελέγχεται στην πολιτική συνοχή, ιδιαίτερα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε επίπεδο ελεγκτικού συνεδρίου. Μέχρι στιγμής ο έλεγχος και από τα διαφθαθεσμικά όργανα επικεντρώνεται σε αμυγός διαδικαστικές ε, έρευνες και οικονομικές σε ό,τι αφορά την ακρίβεια εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και την ε, τακτικότητά τους. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεκτικό Συνέδριο είναι πολύ πιο σημαντικό να μάθουν αν ε, κάποιο πρόγραμμα υπέστη τη σωστή διαδικασία προκήρυξης ε, για, για υποβολή ενδιαφέροντος ή για τον ε, διαγωνισμό και αν τηρήθηκαν οι προθεσμίες. Περισσότερο αυτό τους ενδιαφέρει αν τηρήθηκαν οι προθεσμίες και οι διαδικασίες παρά αν το πρόγραμμα κατέληξε στην κατασκευή των υποδομών για το οποίο προοριζόταν. Αν πραγματικά έγινε ένας αυτοκινητόδρομος, αν πραγματικά δημιουργήθηκε μια γέφυρα, αυτό θα πρέπει να ενδιαφέρει το αποτέλεσμα του προγράμματος και όχι η ευλαβική τήρηση κάποιων διαδικασιών που φαίνεται ότι απασχολεί περισσότερο αυτή τη στιγμή το Ελεκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει στα πλαίσια της διαχείρισης της πολιτικής συνοχής να υποβληθεί και ο στόχος του ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεκτικού Συνεδρίου. Θα πρέπει στα πλαίσια του ελέγχου να, να ελέγχεται και το αποτέλεσμα του προγράμματος και να ελέγχεται και η ίδια η αποτελεσματικότητα του ελέγχου να μην επικεντρώνεται μόνο στις διαδικασίες και να μην εξετάζεται κατά πόσο έγιναν όλα διαδικαστικώς ορθά. Θα πρέπει να δούμε και την ουσία, γιατί το κοινοτικό δίκαιο, οι κοινοτικές διαδικασίες σε μεγάλο βαθμό εφαρμόζονται και εκτελούνται. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα στην εφαρμογή των διαδικασιών. Θα μπορούσαμε επίσης να μιλήσουμε και για πολύ συγκεκριμένες και επιμέρους προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα διεξοδικά να αναλύσουμε κάθε μεμονωμένη πρόταση. Και μάλιστα φαντάζομαι ότι σε πολλές περιπτώσεις ε, θα εξετάσετε όλες αυτές τις προτάσεις στην ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε τώρα. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας τη δική μου παρέμβαση να μιλήσω για ορισμένε πτυχές του νέου δημοσιονομικού κανονισμού που κατά τη γνώμη μας δεν συνάδουν με την απλώστευση, αλλά αντίθετα μεταφέρουν το άχθος του ελέγχου στα κράτη-μέλη και παρά τα φαινόμενα, αντί να πλουστεύει την κατάσταση, την επιβαρύνει και την περιπλέκει ακόμη περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο εκπρόσωπος από την Τσεχία. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, αγαπητά μέλη τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη, καταρχήν θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για τη δυνατότητα που μου δώσατε μαζί με του εκπροσώπου από τη Ζεχία και την Πολωνία, από την ασκοτή και την Πολωνία, να εκπροσωπήσω και εγώ την Τσεχία, το Τσεχικό Υπουργείο Οικονομικών. Να σας πω ότι στα πλαίσια του Υπουργείου είμαι υπεύθυνο αφενός για την πιστοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και αφετέρου για την ετήσια πιστοποίηση της, ε, του αρμόδιου φορέα πληρωμής για τη Γεωργία και ελπίζω ότι με τις ιδιότητες αυτές θα μπορέσω να συγκρίνω την πρακτική εφαρμογή και των δύο συστημάτων, της γεωργίας και της συνοχής και των ε, αντίστοιχων διαδικασιών στα πλαίσια του εθνικού επίπεδου. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε συνοπτικά ότι τα διαρθρωτικά ταμεία ε, συνεργάζονται με τις ε, διαχειριστικές αρχές, τις πιστοποιητικές αρχές και τις ελεκτικές αρχές. Με τρεις βασικούς φορείς δηλαδή. Φυσικά η διαχειριστική αρχή ασχολείται με τη διαχείριση και την εκτέλεση του προγράμματος με βάση τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αντιλαμβάνομαι ότι η αρχή επιστοποίησης ε, σχεδιάστηκε προκειμένου να εξασφαλίσει τα εχέγγια της ε, σωστής διαχείρισης και του ελέγχου και φυσικά οι ελεκτικές αρχές επαληθεύουν κατά πόσο εφαρμόστηκαν σωστά τα, η διαχείριση, τα ελεκτικά συστήματα και διενεργεί και κάποιους ε, δειγματοληπτικούς ελέγχους για την επαλήθευση των δαπανών. Φυσικά υπάρχουν πολλές δυσκολίες στην προσπάθεια συντονισμού του έργου της αρχής πιστοποίησης αφενός και της ελεγκτικής αρχής αφετέρου. Και μερικές φορές λαμβάνουμε κάποιες πληροφορίες για τα σταλίες ή πόνιες απάτης και ως αρχή πιστοποίησης είμαστε υποχρεωμένοι να, να λάβουμε δράση. Βέβαια, με βάση τι κατευθυντήρε γραμμέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να ελέγξουμε επιτόπου κάποια σχέδια και προγράμματα. Το μόνο αποτελεσματικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητήσουμε από του αρμοδίου τη ελεγκτική αρχή να διενεργήσουν του ελέγχου. Και το επιχείρημά του στην αρχή τη περίοδου προγραμματισμού είναι ότι αδυνατούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί εμεί πραγματοποιούμε μόνο δειγματοληπτικού ελέγχου, στι πιστοποιημένε δαπάνε. Πρόκειται για ένα κλειστό κύκλο δηλαδή και από πρακτικής απόψεως ε, καταφέραμε να υπερκεράσουμε αυτό το κόλλημα, αλλά από νομοθετική απόψεως δεν υπάρχει δυνατότητα σε εφαρμογής. Σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, και έχουμε τέσσερι βασικού παράγοντε, τον φορέα πληρωμή, τη συντονιστική αρχή, τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και την αρχή πιστοποίηση. Εδώ έχουμε διαφορετική ορολογία. Ο φορέας ε, πληρωμής έχει παρόμοιες αρμοδιότητες με αυτές της διαχειριστικής αρχής στην, στα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτός ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος. Υπάρχει και μια άλλη υποχρέωση. Τα κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει, μερικά κράτη-μέλη έχουν περισσότερο από έναν φορέα πληρωμής. Οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει μία συντονιστική αρχή, ακόμη και αν υπάρχουν περισσότεροι φορείς πληρωμής, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο σημείο επαφή για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύτερη εναρμόνιση. Υπάρχει τώρα και αρμόδια αρχή. εκεί προβαίνουμε στην πιστοποίηση των φορέων πληρωμής και εξασφαλίζουμε την, εκπλήρωση των κριτηρίων εκ μέρους της, των φορέων πληρωμής και των φορέων πιστοποίησης η αρμόδια αρχή της γεωργικής πολιτικής μοιάζει με την ε, αρχή πιστοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων. Έχουμε και τον τέταρτο φορέα της γεωργικής πολιτικής, το φορέα πιστοποίησης που εξασφαλίζει διεξοδικούς ελέγχους και μάλιστα πιστοποιεί την αλήθεια, πληρότητα και ορθότητα των ε, δαπανών που έχουν πιστοποιηθεί για τους φορείς πληρωμής. Προσπαθώντας να συγκρίνουμε το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προβληματιστούμε με την εξής ερώτηση. Γιατί, για παράδειγμα, την αρχή πιστοποίηση στα διαρθρωτικά μέτρα, τη λέμε έτσι, ενώ ε, στην γεωρική πολιτική η αρχή έχει ελεκτικές αρμοδιότητες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια συνοχή και μια συνέπεια μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της Ένωσης να μην υπάρχουν αποκλήσει. Επίσης, ε, θα πρέπει να διαρωτηθούμε ποιο είναι ο καλύτερο μηχανισμός για να δώσει περισσότερα ειχέγγυα στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εύκολο να διατυπωθεί αυτή η ερώτηση, αλλά δύσκολο να βρεθεί μια απάντηση. Ούτε και εγώ μέχρι στιγμή έχω αποκρισταλώσει τη γνώμη μου για το ποια είναι η ιδανικότερη λύση. Ένας μηχανισμός διαρθρωτικών ταμείων δεν ξέρω αν θα μπορούσε να εφαρμόσει τις άμεσες πληρωμές στη Γεωργία με το ίδιο επίπεδο ελέγχου που ισχύει στο σύστημα διαχείρισης της Γεωργίας. Οπότε είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τις δύο πολιτικές γιατί διαφέρουν. Εν κατακλείδη θα ήθελα να υποβάλω κάποιες προτάσεις για τη μελλοντική συζήτηση που αφορά την απλούστευση της πολιτικής συνοχής θα πρότεινα μια πιο συνεπή και εναρμονισμένη ορολογία για όλες τις πολιτικές. Για παράδειγμα, θα ήθελα να ζητήσω από τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις να, να συντονίζονται καλύτερα μεταξύ τους για μεθοδολογικά θέματα και θέματα ερμηνεών σε όλες τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που ανέφερε και προλαλήσαντες θα πρέπει να αναπτυχθούν κάποιε μεθοδολογίε και να δίδονται στα κράτη-μέλη στην αρχή τη περίοδου για να αποφεύγονται δυσάρεστε εκπλήξει στα μέσα τη περίοδου προγραμματισμού. Γιατί τότε είναι δύσκολη η αντίδραση. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια τη επιλεξιμότητα, πιστεύω ότι τα κριτήρια που καθορίζουν οι κανονισμοί θα πρέπει να ισχύουν για όλε τι πολιτικέ. ΦΠΑ, για παράδειγμα διαφορετική διαχείριση του ΦΠΑ παρατηρούμε στα διαρθρωτικά ταμεία και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Συμφωνώ με τον Γκράχαμ σε πολλά σημεία. Πιστεύω ότι η απλούστευση των μηχανισμών ε, εκτέλεσης θα πρέπει να γίνεται με εξέλιξη περισσότερο παρά με παραστατικές μεθόδους και επίση ε, να αξιοποιήσουμε την παρούσα κατάσταση, παρόλο που υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Έχω την αίσθηση ότι οι νέε χώρε μέλη έχουν αρχέ πιστοποίησης πολύ καλά στελεχωμένες, που δίνουν περισσότερα εχέγγυα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κρατη για τη σωστή διαχείριση. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι οι χώρες του Βίσεγκρατ θα εκπονήσουν κοινό έγγραφο για τους μηχανισμούς καλύτερης εφαρμογής της πολιτικής συνοχής και θα υποβάλουμε το κοινό μας αυτό έγγραφο προς το τέλος του έτους και στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Γκρέγκορ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συμμετέχοντες για ερωτήσεις, για σχόλια. Ο κύριος Σρέντερ. Η κυρία Σρέντερ. Το πρώτο μου σχόλιο. Είναι ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Είμαι αρκετά απογοητευμένη που οι εμπειρογνώμονες δεν κάνουν καμία συγκεκριμένη πρόταση. Γνωρίζουμε την κατάσταση, σε εν πάση λεπτομερία θα έλεγα. Και ξέρουμε πολύ καλά γιατί ε, τα πράγματα φτάσανε όπου φτάσανε, σε αυτό το αδιέξοδο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ελεγκτικό συνέδριο ε, ψάχνει πολύ περισσότερα τα πράγματα τώρα, γιατί υπάρχουν προβλήματα με την εφαρμογή των κονδυλίων των διαφορετικών ταμείων. Αλλά το δικό μας το ερώτημα ήταν κάτι διαφορετικό. Θέλω μια αξιολόγηση με βάση τα αποτελέσματα για να ξεπεράσουμε, αυτό το επίπεδο, να ξεπεράσουμε το επίπεδο του ελεγκτικού συνεδρίου και να δούμε τι κάνουμε μετά. Ξαναθέτω το ερώτημα στους εμπειρογνώμονες. Γιατί δεν κάνουμε έναν έλεγχο ανάλογα με τα αποτελέσματα. Ε, μιλάμε για δημόσια χρήματα. Έχουμε καθήκον απέναντι στους φορολογούμενους να τα σωστά. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ο έλεγχος δεν είναι απλώς ε, διαδικαστικός. Πώς ε, θα εξασφαλίσουμε ότι δίνει και αποτελέσματα. Πώς θα εξασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια ξοδεύονται με ακρίβεια, με διαφάνεια και επιτρέπει στους φορολογούμενους να γνωρίζουν γιατί πληρώνουν, πού ξοδεύονται οι φόροι τους. Αυτή είναι η απάντηση που θέλουμε. Η ανάλυση σα ήταν ενδιαφέρουσα, αλλά δεν μας είπε τίποτα καινούριο, τίποτα που να μην ξέρουμε. Ο κύριος Φανίστελ Ρόι. Οι πληροφορίε ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα. Μιλάτε για μια εξέλιξη και όχι για μια επανάσταση. Ωραία, αλλά προς ποια κατεύθυνση θα γίνει αυτή η εξέλιξη. Η εξέλιξη. Τώρα θα αναθεωρήσουμε το γενικό δημοσιονομικό κανονισμό των ταμείων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι όλα τα ταμεία που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, σε επίπεδο εκτέλεση στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να υποστούν ένα εξορθολογισμό, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ευθύνες του καθενός, να είναι σαφώς οριοθετημένες. Συνήθως αυτές οι ευθύνε είναι σε επίπεδο κράτους μέλους. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Μας είπατε ότι αυτή η δήλωση αξιοπιστίας των κρατών μελών θα πρέπει να είναι πολύ πιο ακριβής από πλευράς κρατών μελών. Αλλά ακούστε, κοιτάξτε, πριν από δύο μήνες το πολύ Μεταβήκαμε στη Γαλλία. Και έγιναν 4 ή 5 έλεγχοι και μετά από 4 χρόνια δεν υπάρχουν αποτελέσματα. Το, το σύστημα είναι απίστευτα περίπλοκο, το εξηγήσαμε, το ξαναεξηγήσαμε 4-5 φορές, αλλά παραμένει περίπλοκο. Όπω είπατε και εσεί δεν πρόκειται περί επανάσταση. Αλλά από τη νέα προγραμματική περίοδο θα πρέπει να υπάρξουν κάποιε αλλαγέ. Προ ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε, λοιπόν. Και όπω είπε και ο τελευταίο ομιλητή. ορισμένοι θεωρούν ότι πρέπει να υιοθετήσουμε τους κανόνες του Γεωργικού Ταμείου. Εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ριζοσπαστικά διαφορετική μέθοδο σε ό,τι αφορά την κατανομή τους ε, και την ε, ροή τους προς τους δικαιούχους. Πώς βλέπετε τα πράγματα. Τι μας χρειάζεται, ένας νέος κανονισμός, τι μας χρειάζεται ακριβώς. Ο Γιάννη Κοσβόφσκι. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία πρόταση που προκύπτει από την εμπειρία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στο άρθρο 39 του Γενικού Κανονισμού θα πρότεινα αυτά τα major projects, τα μείζωνα σχέδια που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια και όχι τα 25 εκατομμύρια για τα περιβαλλοντικά προγράμματα και 50 για τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι έτσι θα πλουστεύσουμε τα πράγματα και για τα κράτη-μέλη αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερη πρότασή μου αφορά την ε, βράχηση της περίοδου ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το άρθρο 57 του Γενικού Κανονισμού. Από τρία να γίνουν δύο χρόνια η προθεσμία, γιατί η τριετής προθεσμία είναι υπερβολικά επιβεριντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και περιορίζει την ανταγωνιστικότητά τους. Προτείνω λοιπόν την περίοδο, τη διετή περίοδο. Σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του ελέγχου, αυτή είναι η τρίτη μου πρόταση, θα πρέπει η διαχείριση να γίνει ενιαία σε κοινοτικό επίπεδο. Από την προσωπική μου πείρα διαπίστωσα ότι μέσα σε ένα μήνα μπορούν να γίνουν διάφορες, διάφοροι έλεγχοι σε, σε διάφορα επίπεδα στην ε, Πολωνία σε τρεις διαφορετικούς ελεκτικούς φορείς, κάτι που επιβαρύνει πολύ τα πράγματα για την ε, χώρα. Να ακούσω άλλα σχόλια. Ε, σχόλια από τους εμπειρογνώμονες ενώ Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να απαντήσει, ας πάρει το λόγο. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Δυστυχώς ε, η απλούστευση ε, είναι η λαθασμένη λέξη, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει μια απλότητα στην όλη διαδικασία. Όπως είπα, στο τέλος παρουσίασής μου, έχουμε ένα απίστευτα περίπλοκο σύστημα επιμερισμένης διαχείρισης. Αν δείτε άλλες αναπτυξιακές οργανώσεις ή άλλα πολυμερή συστήματα, βλέπουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες προκλήσεις στα κράτη-μέλη. Το σύστημα διαχείρισης σε πολλά επίπεδο τουλάχιστον έχει ένα πλαίσιο, το κρατικό. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 κράτη-μέλη και κάθε κράτος μέλος με διαφορετικό θεσμικό ας πούμε, χαρακτήρα, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ε, ένα απλό σύστημα θα ήταν απλώς μεταφορές ε, από τον προϋπολογισμό από το ευρωπαϊκό επίπεδο στο εθνικό επίπεδο. Αλλά προσπαθούμε να έχουμε όμω και πολιτική συνοχή. Έτσι δεν θα είχαμε πολιτική συνοχή. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή σα και την ενόχλησή σα. Η λύση δεν είναι, κατά γνώμη μου, στην εξέβρεση μιας μαγικής λύσης. Αλλά διάφορες από τις παρουσιάσεις που ακούσατε σας δείχνουν με πολύ καλό τρόπο ε, τι θα μπορούσε να γίνει, ε, κάποια θετικά βήματα που θα μπορούσαν να προωθηθούν. Ο Γιάνν Γκρέγκο συνόψισε αυτό που είπαμε πολύ, εμπειρογνώμονες. Ήρθε κανόνες επιλεξιμότητας, ε, συνεπείς μεθοδολογίες, σταθερότητα των κανόνων, πριν και κατά τη διάρκεια περίοδο του προγραμματισμού, ε, συνεκτική προσέγγιση Στου ελέγχου. Άλλο απάτη, άλλο άλλες παρατυπίες. Να τις διαχωρίσουμε. Είναι πρακτικές συστάσεις νομίζω αυτές που είναι ένα πρακτικό εργαλείο για να προχωρήσουμε. Νομίζω, αν τι ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μπάχλερ. Άλλος κανείς από τους εμπειρογνώμονες θα ήθελε να απαντήσει. Για τις ερωτήσεις του κυρίου Βανίστελ Ρόι να απαντήσω. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε με τον χρηματοδοτικό κανονισμό. Ε, δύσκολο ερώτημα, δύσκολη απάντηση. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να βασιστούμε στα εθνικά συστήματα διαχείρισης και ελέγχου. Στην Τσεχία, παραδείγματο χάρη, έχουμε τρεις φορείς ε, στη διαχείριση και τον έλεγχο των εθνικών κονδυλίων ένας ε, αξιωματούχος ε, έγκρισης, ένας διαχειριστής και ένας λογιστής. Οι ίδιοι κανόνες υπάρχουν και στην Κομισιόν. Υπάρχει ο αξιωματούχος που είναι ο διατάκτης και ο λογιστής. Μπορούμε να βασιστούμε στα εθνικά συστήματα ελέγχου, να τα σεβαστούμε και να μην ε, βάλουμε κι άλλα στρώματα για την, ε, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες. Γιατί αυτό ο διαχωρισμό που έχουμε κάνει, ε, διαχειριστική αρχή, αρχή επιστοποίηση και αρχή ελέγχου, είναι λίγο τεχνητή. Παραδείγματο χάρη, στην αρχή διαχείριση. Κρατάμε αυτέ τι τρει λειτουργίε που έχουμε σε εθνικό επίπεδο. Διατάκτη, υπάλληλο προπολογισμού και πώς ένα... Και ο ελεγκτή είναι ο τρίτος. Επομένως, λοιπόν, να σεβαστούμε το εθνικό σύστημα, την εθνική διαστρωμάτωση. Και εγώ έχω ένα σχόλιο. Όπως είπε ο καθηγητής Μπάχτλερ, ίσως θα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο μέτρο ε, να μεταφερθούν ε, οι αρμοδιότητες ε, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Φυσικά θα υπάρξουν παρατυπίες, ατασταλίες, σφάλματα γίνονται, αλλά έτσι θα, γίνονται, θα γίνουν ρηξικέλευθες αλλαγές στο σύστημα. Και αν εσείς πιστεύετε ότι αισθάνεστε μηχανία και απογοήτευση, εκνευρισμό, φανταστείτε ε, τους ετούντες που είδαν τόσες πολλές αλλαγές στα διάφορα συστήματα, στις προγραμματικές περίοδου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που υποβάλλουν ε, τις αιτήσει τους και θα πρέπει οι διαχειριστικές αρχές να ε, ικανοποιήσουν τις, ε, τους 8 διαφορετικούς ελέγχους μέσα σε ελάχιστες προθεσμίες και αισθάνονται ότι βρίσκονται χαμένοι στο σκοτάδι, είναι τελείως αβοήθητοι και κάνουν ό,τι μπορούν για τη σωστή διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων. Και είναι αδύναμοι οι μηχανισμοί ελέγχου. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάποια διεθνή κριτήρια και προδιαγραφέ, αυτά να σεβαστούμε, ε, να τα εφαρμόσουμε παντού και έτσι θα έχουμε τεράστιες αλλαγέ και στα συστήματα διαχείρισης και στα συστήματα ελέγχου σε όλα τα διαρθρωτικά ταμεία. Ο κύριο ε, Καρου, Καλούπα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ερώτηση πώς θα αναγνωρίσουμε την αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου και του Ελεκτικού Συνεδρίου σε ό,τι αφορά την ετήσια καθάριση λογαριασμών. Φάνηκε από αυτά που είπαμε ότι και στι αρμοδιότητες του Ελεκτικού Συνεδρίου και στι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπάρχουν, τερά, υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες γιατί μέχρι στιγμής ε, ε, υπάρχουν πολλά κριτήρια διασταυρωμένα και η τήρηση των διαδικασιών είναι πολύ δύσκολη. Και αν δεν προκαθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες του ελέγχου και αν δεν ε, επικεντρωθούν οι έλεγχοι στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής, στην ουσία δηλαδή, και ξεφύγουν από τις διαδικασίες και την ευλαβική τους ε, τήρηση, τότε δεν θα έχουμε πραγματική πρόοδο. Και είναι κάπως τεχνητό το όριο των 2%. Επαναλαμβάνω, προσπαθούμε να, να θεραπεύσουμε κάποια συμπτώματα, αλλά η αιτία μένει θεράπευτη. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και όχι μόνο των διαδικασιών της πολιτικής συνοχής. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Κυρία Σάντζες Σμιθ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα πολύ προσεκτικά τους εμπειρογνώμονες και έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πρόβλημα μεταξύ του στόχου της απλούστευσης και της ανάγκης ε, ε, του περιορισμού των σφαλμάτων και της πιο αυστηρής εφαρμογής. Απ' τη μια θέλουμε να εκλεπτύνουμε τον έλεγχο και απ' την άλλη να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Και μάλιστα η απλούστευση στην περίοδο 2001-2006 προκάλεσε αντιδράσεις σφοδρές στα κράτη-μέλη και ένας εμπειρογνώμενος μας είπε ότι είναι πολύ δύσκολο στην πορεία να αλλάξουν τα πράγματα, όπως συζητήθηκε από την πρώτη προγραμματική περίοδο. Θέλουμε λοιπόν λιγότερες ε, διοικητικές απαιτήσει, μεγαλύτερη διαφάνεια και όλοι για να είναι ε, σωστοί απέναντι στο ελεκτικό συνέδριο θέλουν να διενεργήσουν τους ελέγχους τους και να περιορίσουν τα σφάλματα. Οπότε αυτές οι τροποποίησεις που έγιναν στην πορεία φυσικά δεν είναι ρήξη και έλευθες, είναι κάποιες αλλαγέ μικρές. Ουσιαστικά πρόκειται για προσαρμογή και όχι για αναθεώρηση. Πώς εφαρμόζονται και επίση. Πότε έγιναν, πότε θεσπίστηκαν οι κανόνες για την τωρινή περίοδο, το 2004. Ε, άρχισαν να ισχύουν το 2007. Σήμερα όμως ε, βρισκόμαστε στο 2010 με κανόνες όμως που θεσπίστηκαν το 2004. Η σημερινή κατάσταση διαφέρει αρκετά από αυτή που επικρατούσε το 2004 όταν πρώτο θεσπίστηκαν αυτοί οι κανόνες. Ας το σκεφτούμε και αυτό. Πώς θα προσαρμόσουμε τους παλιούς κανόνες στη σημερινή κατάσταση. Ίσως ε, ο κανονισμός αυτός, επειδή ακριβώς καταρτίστηκε σε προηγούμενη περίοδο, δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες. Σε ό,τι αφορά το περιθώριο λάθους, υπάρχουν καλοί και λιγότερο καλοί μαθητές στις χώρες μέλη. Ίσως οι λιγότερο καλοί μαθητές θα πρέπει να διορθώσουν τα λάθη τους και θα πρέπει να βοηθήσουν αυτές τις χώρες για να διορθώσουν τα περιθώρια λάθους. Οι χώρες όμως που έχουν καλύτερες επιδόσεις δεν θα πρέπει να επιβραβευθούν με μια ελάφρυση των ελέγχων, ίσως να συναυθούν κάποιες συμφωνίες εμπιστοσύνη, ε, συμβόλαια εμπιστοσύνη μαζί τους. Συμφωνώ με τις κυρώσεις για τις χώρες που έχουν μεγάλο περιθώριο λάθους, αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να βελτιώσουν τους ελέγχους τους και να περιορίσουν το περιθώριο λαθών τους. Ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Έχω να σας κάνω μια πρόταση, γιατί ε, προσωπικά δυσκολεύομαι να καταλάβω ορισμένα πράγματα. Και η πρόταση που έχω να σας κάνω, κυρία Πρόεδρε, είναι η εξή. Αν μπορούν οι αξιότιμοι εισηγητέ να κάτσουν γύρω από ένα τραπέζι και να μας φέρουν ένα χαρτί με τις φωτάσεις τους. Και θα σας πω γιατί. Από πολλούς τελικά η συζήτηση οδηγείται στο θέμα ασφάλματα ή απάτη. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σωστό και πολύ καλά ότι αυτό το ζήτημα τέθηκε και δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι τέθηκε καταρχήν από τον κύριο που εκπροσωπεί την κυβέρνηση της Πολωνίας, νομίζω και από τον κύριο από την ε, Τσεχία. Και συζητάμε για ένα θέμα το οποίο δεν ήταν καν αντικείμενο της μελέτης. Ούτε στη μελέτη του κυρίου Μπάτσλερ υπάρχει το ζήτημα, και ούτε στην άλλη μελέτη έχουμε το οποιοδήποτε στοιχείο για το πώς η διαδικασία απλούστευσης έχει επηρεάσει τις απάτες και τα σφάλματα. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Δεν ξέρω γιατί τέθηκε αυτό το θέμα, καλώς τέθηκε. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει ένα πρόβλημα με το τι συζητάμε. Ε, προέρχομαι από μια χώρα που το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, όπως είναι γνωστό, δεν έχω καμία δυσκολία να το πω. Όμως, εφόσον συζητάμε για διαδικασία απλούστευσης, πρέπει να ξέρουμε και τι ζητάμε. Δεύτερη, ε, δεύτερο ζήτημα που ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που σας πρότεινα. Παραδείγματο χάρη, στην, ε, στην μελέτη του κυρίου Μπάτσλερ, ε, είναι ο πίνακας, ο κάθετος με τα τρία χρώματα, το κίτρινο, το κόκκινο και το μπλε όπου φαίνεται ότι τα μέτρα ήταν καλά μέχρι πολύ καλά της απλούστευσης. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα εγώ. Στη μελέτη ε, του κυρίου ε, Μπλόμεγε Σάντσες και σας παραπέμπτω στη σελίδα μισό λεπτό τη βρω σελίδα ε, μισό λεπτό εδώ βρίσκω εδώ στη σελίδα 8 και 9 ειδικά στη σελίδα 9, 71% αυτών που απαντάν μας λένε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές σημαντικές στο θέμα της, ε, της απορρόφησης ας πούμε. Ή αν πάμε στην προηγούμενη σελίδα θα δούμε ένα 60% βλέπουν ότι οι ε, administrative επιβαρύνσεις δεν έχουν αλλάξει. Αναρωτιέμαι τώρα, μεταξύ των δύο μελετών, ποια είναι η σωστή, ποια μου δίνει εμένα τα, καλά, τα σωστά συμπεράσματα. Τρίτο ζήτημα και τελειώνω με αυτό. Θεωρώ πράγματι ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα που έθεξε ο κύριος ε, Μπάτσλερ όσον αφορά το ρίσκο. Σε σελίδα 13 όπου θέτει το ερώτημα ποια είναι τα αποδεκτά ρίσκα για την ε, πολιτικής συνοχής χωρίς όμως να απαντάει και χωρί να μας δίνει και κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε αυτά τα, να υπολογίσουμε αυτά τα ρίσκα και φυσικά υπάρχει στην, στην ίδια σελίδα η πρόταση ή σκέψη του κυρίου για το θέμα της εναρμόνισης των κριτηρίων επιλεξιμότητας Αυτέ όμω είναι, ειδικά αυτή η πρόταση, είναι μια τυπική πρόταση. Ο καθένα καταλαβαίνει ότι αν είναι ενιαία τα κριτήρια επιλεξιμότητα, προφανώ θα είναι και πιο εύκολη η διαδικασία διαχείριση των έργων. Αλλά μια τέτοια πρόταση έχει ορισμένες, ορισμένα μειονεκτήματα, τα οποία καλό είναι να παθούν υπόψη. Τέλο, και εγώ νομίζω ότι τελικά αυτό που πρέπει να μα απασχολεί είναι αυτό που είπε ο, να με συγχωρεί ο κύριο ε, εκπρόσωπο από την Πολωνία, δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν είναι διαδικασίε. Και εγώ πιστεύω ότι οι διαδικασίε είναι σωστέ εμπολή. Το πρόβλημα είναι εάν ένα ποσό για κάποιο έργο οδήγησε στην υλοποίηση του έργου και όχι. Ή όχι. Ή με ποια ποιότητα. Και γι' αυτό το θέμα δεν έχουμε καμία διαδικασία αξιολόγηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Uh, dear colleagues, we still have... Αγαπητοί συνάδελφοι, τρεις συνάδελφοι ζητούν το λόγο και μετά θα πρέπει και η Κομισιόν να μιλήσει. Οπότε ας είμαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι και παρακαλώ αναφέρετε σε ποιον απευθύνεται το ερώτημα. Γιάνν Ολμπριχτ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Ε, ε, I Καταρχήν να ευχαριστήσω για τις πληροφορίες και την έρευνα. Βέβαια οι εμπειρογνώμονες δεν μπορούν να μας δώσουν λεπτομερείς προτάσεις. Οι προτάσεις είναι απόρρια αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν. Δεν μπορεί να προηγούνται οι προτάσεις των αποφάσεων. Στο Κοινοβούλιο νομίζω ότι έχουμε το εξής, την εξής ενδιαφέρουσα κατάσταση. Στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών γίνεται η συζήτηση με το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο επικρίνει την ε, Κομισιόν για κάποια σφάλματα. Τα μέλη του Κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου μπερδεύουν σφάλματα με απάτες και συζητούμε για το πιθανό επίπεδο σφαλμάτων παρόλα αυτά, το ελεγκτικό συνέδριο ζητεί ουσιαστικά περισσότερους ελέγχους από την Κομισιόν. Ταυτόχρονα έχουμε το πρόγραμμα ανάκαμψης και συζητούμε και για την απλούστευση. Όλα αυτά ταυτόχρονα. Πώς θα απλουστεύσουμε κάτι ενώ απαιτείται αυξημένος έλεγχος. Ταυτόχρονα συζητούμε για το δημοσιονομικό κανονισμό και έχουμε επιτάπητος, όπως ξέρουν τα μέλη της Επιτροπής αυτής, Έχουμε τις πρώτες προτάσεις από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού για το πώς θα συνδυάσουμε τις διαδικασίες από την Άγκρη και τα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι, υπάρχουν, έχουν κατατεθεί προτάσεις. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές, τελείως διαφορετικές πολιτικές. Πώς θα γίνει. Αυτό που χρειαζόμαστε και φαίνεται από αυτό που είπαν οι εμπειρογνώμονες είναι να επιλέξουμε δύο στρατηγικές εξελικτική η μία. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι που είναι περίπλοκο, αλλά σε 10-15 χρόνια θα τα καταφέρουμε. Ή πιο εξελικτικά, πιο επαναστατικά. Να θέσουμε το ερώτημα πώς ορίζομαι την επιμερισμένη διαχείριση. Επιμερισμένη διαχείριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με 27 διαφορετικά συστήματα και να έχουμε ένα επιμερισμένο. Το κέριο ερώτημα είναι το ζήτημα της επιλεξιμότητας. Θα πρέπει να έχουμε εναρμονισμένα κριτήρια επιλεξιμότητα σε όλες τις επενδύσεις ή θα έχουμε επιλεξιμότητα για το ευρωπαϊκό κομμάτι και άλλο σύστημα επιλεξιμότητας για το εθνικό κομμάτι που είναι τα δύο αντιφατικά και εκεί πια χάνονται μέσα στα συστήματα και οι δικαιούχοι. Θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη. Όχι να τους στέλνουμε τα χρήματα, να τους τα εμβάζουμε, αλλά να καθιστούμε τα κράτη-μέλη υπεύθυνα για την υλοποίηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο. Ή δεν θα εμπιστευτούμε τα κράτη-μέλη λόγω των προσφαλμάτων κλπ. Και θα τους δώσουμε την δυνατότητα, ελέγχοντάς τα όλο και περισσότερο. Τι θα κάνουμε λοιπόν, είτε θα δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη, ίσως ε, αργότερα θα επαληθεύουμε αυτά που μας λένε. Αλλά αν έχουμε δύο κέντρα λήψης αποφάσεων, θα μπερδευτούμε. Δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε ολόκληρο το σύστημα της ε, ε, κατανομής των κονδυλίων, γιατί υπάρχουν διαφορές στα συστήματα. Στον γεωργικό τομέα δεν έχουμε ε, το σύστημα των διαγωνισμών. Και στα διαφορετικά ταμεία έχουμε 27 διαφορετικά συστήματα. Άρα το κέριο ερώτημα είναι πώς ορίζουμε την επιμερισμένη διαχείριση. Και αν δούμε σοβαρά το θέμα, τι πρέπει να εναρμονιστεί. Οι κρατικές προμήθειες, η επιλεξιμότητα, και ποια είναι η πραγματική ευθύνη των κρατών μελών. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε μεγαλύτερη περιπλοκότητα, αυξημένους ελέγχους και η όλη ευθύνη θα ανατίθεται στα κράτη-μέλη χωρίς τα κράτη-μέλη να έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις. Τα κράτη-μέλη δηλαδή θα αυξήσουν τους ελέγχους, θα ε, τους επιβάλλουν στους ε, αποδέκτες, οι οποίοι θα εξοργιστούν και θα έχουμε βλέπουμε ότι έχουμε πολλούς ε, δυνάμει δικαιούχους που παρατούνται από τη δυνατότητα αξιοποίησης ε, κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάνε να πάρουν δάνειο από τις τράπεζες γιατί λένε ευχαριστώ πολύ, πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε πολιτικές αποφάσεις, μετά θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες και θα πρέπει να συζητήσουμε και τις εθνικές δηλώσεις και ε, θέματα αξιοπιστίας, ασφάλισης αλλά Είτε θα δείξουμε εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη, όπως είπα, και θα παίρνουμε τις πληροφορίες για το πώς εξελίσσεται το πρόγραμμα ή όχι και θα τα κάνουμε όλα συγκεντρωτικά στις Βρυξέλλες. Αλλά νομίζω ότι αυτό το σύστημα δεν θα μας πάει μακριά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που μας είπε προηγουμένως ο κύριος Όλμπριχτ. Θα ήθελα να προσθέσω ορισμένα πράγματα όσο πιο απλά και κατανοητά γίνεται. Κατά τη γνώμη μου, απλούστευση θα πρέπει να σημαίνει ένα σύστημα πιο εύληπτο, πιο κατανοητό και χρειαζόμαστε και συνεπιορολογία και εναρμονισμένη μεθοδολογία και για τους ε, διαγωνισμούς, να έχουμε στο μέτρο του δυνατού παρόμοια κριτήρια επιλογής ή επιλεξιμότητας. Δεν μπορούμε το ΦΠΑ να τον περιλαμβάνουμε μόνο σε ένα ταμείο και όχι στα άλλα. Θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. για την έγκριση των σχεδίων και στα κράτη-μέλη και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης τα ίδια κριτήρια να ισχύουν και για την πληρωμή. Όλοι αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να είναι σταθεροί, να μην αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο, για να μην αποθαρρύνονται οι ετούντες, ιδιαίτερα όταν δεν είναι πολυεθνικές. Ε, ευχαριστώ. Ότι πέσαμε σε μία παγίδα. Γιατί α, ελέγχουμε τα προγράμματα, ενώ αυτό που θέλουμε να δούμε ε, είναι αν ξοδεύουμε τα λεφτά ε, για αυτό που τα ζητήσαμε. Ακούσαμε μία φράση, δύο φράσεις, ε, από τον Πολωνό συνάδελφο που είπε «Κανένας δεν μας ρώτησε αν χτίστηκε η γέφυρα, ας πούμε». Πολύ ομιλούς αυτή η εικόνα. Οι Σκοτσέζοι είναι γνωστοί για τη ζυγκουνιά τους. Ε, και γι' αυτό έχουμε πάρει μάλλον λάθος τροχιά. Ορισμένα προγράμματα του κοινωνικού ταμείου δεν υλοποιούσαν τους στόχους που είχαν καθοριστεί από την αρχή. Κάτι χάνουμε εδώ πέρα, χάνουμε το στόχο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάποιοι αξιωματούχοι που θα ελέγχουν κάτι σε επιθεωρήσεις για να δούμε αν υπάρχουν, αν εξελίξει και τρέχουν τα προγράμματα, αν όχι, να διδαχθούμε από αυτό, να βοηθήσουμε αυτούς που προσπαθούν να υλοποιήσουν τα προγράμματα για τα οποία ζήτησα χρηματοδότηση, να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να είναι επιτυχημένα. Πρέπει να είμαι σε θέση να λέμε στους πολίτες τα κονδύλια σας ε, ξοδεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο και μικροί επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να γίνονται είτε από εδώ είτε να πηγαίνουν κάποιες ε, μικρές ομάδες επιτόπου αλλά χρειαζόμαστε μια αξιολόγηση προγραμμάτων και όχι να πηγαίνουν αυτοί που μετράνε τα κουκιά ας πούμε, και τσακίζουν τον κόσμο με τις ερωτήσεις. Ας πούμε. Γιατί αλλιώς απλώς θα αποθαρρυνθεί ο κόσμος να μην κάνει αιτήσει, ας πούμε. Και αυτό ε, είναι, θα ήταν απαράδεκτο, θα ήταν κρίμα. Ε, κυρία Χίμπνερ, ε, ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα προς εσάς και προς την ε, Κομισιόν. Ξέρετε ότι την Κομισιόν πριν από λίγο ολοκλήρωσε την αξιολόγηση συμμόρφωσης. Και λίγο πολύ όλα τα κράτη-μέλη έχουν λάβει αυτές τις αξιολογήσεις. Πριν να Έχουμε άλλα τρία χρόνια πριν την νέα προγραμματική περίοδο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης ως εγγύηση για την επόμενη για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Να μην ξανακάνουμε δηλαδή τέτοιες αξιολογήσεις, αλλά να έχουμε συστήματα όπου αυτές οι αξιολογήσεις που έχουν ήδη γίνει σε ένα κράτος μέλος να αποτελέσουν τη βάση και για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Τώρα, όποιο θέλει να απαντήσει, η Κομισιόν ή οποιο έχει να πει κάποια καταληκτικά λόγια, δεν ξέρω ποιο θέλει να ξεκινήσει. Θα απαντήσω το εύκολο για τη συμμόρφωση. Πιστεύω ότι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης είναι καθημερινή δουλειά. Η Κομισιόν θα πρέπει να δεχτεί τα περιεχόμενα, θα κριθεί με βάση αυτά και θα τα χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε μελλοντικό πρόγραμμα για την περίοδο 2007-2013. Τώρα, αν αλλάξουν μετά άρδιν τα πράγματα, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Είναι καλή βάση. Οποια... Βέβαια, οποιασδήποτε μίζονες αλλαγές θα απαιτήσουν και μίζονες άλλες αλλαγές ε, από την πλευρά των κρατών μελών. Για να απαντήσω στην ερώτηση από τον Έλληνα ε, συνάδελφο του οποίου το όνομα δυστυχώς δεν συγκράτησα για τις έρευνες και την αποτελεσματικότητα των μέτρων, νομίζω ότι γενικά μπορούμε να πούμε ότι είναι νωρίς, είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε ε, αξιόπιστα την αποτελεσματικότητα των μέτρων γιατί είναι πολύ εξειδικευμένα πολλές φορές και είναι δύσκολο να κρίνουμε τον αντίκτυπο που θα έχουν για παράδειγμα στο ποσοστό σφαλμάτων. Υπάρχουν διαφορές όντως μεταξύ των ε, ε, ερευνών. Μπλόμαϊερ και δικών μας λόγω της διαφορετικής μεθοδολογίας διαφορετικών ερωτήσεων που ετέθησαν και απαντήθηκαν. Ε, το ένα αφορούσε τη γνώμη των διαχειριστικών αρχών, η άλλη των αρχών ελέγχου. Και υπάρχουν διαφορές ενδεχομένως μεταξύ το, της γνώμης των δύο. Επίσης υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ επιμέρους μέτρων. Αν θέλει κανείς να δει θέματα αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να δει το συγκεκριμένο μέτρο. Ο Γκραμ Βάτσον είπε κάτι σχετικά. Πολλά μέτρα είχαν θετικό αντίκτυπο για πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες όμως ε, στην διοίκηση και μπορεί να μην μειώσουν συνολικά το διαχειριστικό ή διοικητικό φόρτο. Επίσης, ε, πολλές διαχειριστικές αρχές ε, αρέσκονται σε καταποκοπήν ποσά. Αυτό όμως χρειάζεται μεγαλύτερη διαχειριστική προσπάθεια και διοικητική προσπάθεια ε, βράχη πρόθεσμα, ούτως ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γκραμ. Θα σχολιάσω δύο πράγματα. Βέβαια, οι παρεμβάσει στα διαρθρωτικά ταμεία και στη γεωργική πολιτική διαφέρουν πολύ. Αλλά από άποψη συστημική νομίζω ότι η γεωργία έχει ένα σύστημα που μπορεί να αντιμετωπίσει τα πολυετή προγράμματα για την ανάπτυξη της υπαίθρου, για παράδειγμα, και το ετήσιο κλείσιμο των λογαριασμών είναι εφικτό. Αλλά είναι διαφορετικό. Τώρα για τη διαπίστευση να πω κάτι. Ε, θα είναι δυνατή για τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Στη γεωργική πολιτική θα πρέπει να διαπιστέψω με βάση τον πλήρη έλεγχο του συστήματος πριν αρχίσουμε. Μετά ε, με βάση τους κανονισμούς στη Γεωργία θα πρέπει να παρακολουθώ συνεχώς ε, τα κριτήρια της διαπίστευσης ε, υπιστοποίησης. Άρα θα πρέπει κάθε τρίμηνο να βλέπω τον οργανισμό πληρωμών και να τσεκάρω ότι όντως πληρούνται όλα τα κριτήρια. Και υπάρχει και η προϋπόθεση για το... την έκθεση τρεις φορές το χρόνο. Ρώτησα τους συναδέλφους από τη Διεύθυνση Γεωργίας τι σημαίνει η διαπίστευση και είπαν ότι θα πρέπει από την αρχή να ακολουθηθεί, να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Οπότε εδώ υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές. Επίσης ο δημοσιονομικός κανονισμός κάπου λέει ότι οποιοδήποτε ρόλος της Κομισιόν μπορεί να ορίζεται από κανονισμούς ειδικού ανατομέα. Και ρωτώ γιατί. Γιατί στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας δέχεται την Εθνική Διαπίστευση Κομισιόν και γιατί στη Γενική Διεύθυνση, γιατί η Γενική Διεύθυνση για την περιφερειακή ανάπτυξη θα πρέπει να ε, ενέχεται σε αυτή τη διαδικασία ε, χορηγώντας έγκριση. Να σχολιάσω δύο σημεία που δεν απαντήθηκαν. Το ένα φέρθηκε στους ελέγχους και τι θα πρέπει να ελέγχεται. Ήμουν και ελέγχτης κάποτε και είναι εύκολο να ελεγχθούν αριθμοί, λογαριασμοί. Αλλά πώς θα ελέγξει ένας ελέγχτης το αποτέλεσμα, αν πραγματικά κατασκευάστηκε η γέφυρα. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει διαφορετική μεθοδολογία, διαφορετική νοοτροπία και διαφορετικό είδος ελέγχου. Γιατί είναι εύκολο να ελεγχθούν αριθμοί, βιβλία, λογαριασμοί, αλλά το αποτέλεσμα για να ελεγχθεί χρειάζεται τροποποίηση της φιλοσοφίας του ελέγχου. Επίσης, σε ό,τι αφορά την συνεργασία της Επιτροπής και της CCA, φαίνεται ότι η CCA ε, ζητά περισσότερους ελέγχους, προσπαθεί να είναι πιο απαιτητική και λέει ότι υπάρχουν πολλοί έλεγχοι. Και αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Έχουμε πολλούς ελέγχους, αλλά πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε την μόνιμη απέτηση του ελεκτικού συνεδρίου για ένα ε, σύστημα που θα είναι και αποτελεσματικό αλλά και θα καλοποιεί τους στόχους με μικρές αλλαγές. Και σε ό,τι αφορά το χαμηλό ποσοστό λάθους που έχουν ορισμένες πολιτικές δεν σημαίνει ότι αν μετα... μεταφερθεί στο... στα διαρθρωτικά ταμεία η μέθοδος αυτή θα περιοριστεί και το περιθώριο ε... λάθους ε, και στα διαρθρωτικά ταμεία. Κύριε Καλούπε θέλετε να προσθέσετε κάτι, όχι, κύριε Μπλομ Μέγερ. Ο Πίτερ Μπέρκοβι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες και τα μέλη της Επιτροπής σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ακούσαμε με προσοχή. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Μπλομάιερ για τη διαβούλευση. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε τις πιο εντατικές διαδικασίες συζητήσεων και διαβουλεύσεων με εμπειρογνώμονες στα κράτη-μέλη και σε περιφερειακό επίπεδο. Και το κάναμε αυτό στη βάση ομάδων εργασιών και άλλων επαθών όμως. Και μας βοήθησε να εντοπίσουμε διάφορα μικροπροβλήματα. Δόθηκε ένα έντονο μήνυμα από τους εμπειρογνώμονες, ε, τα κράτη-μέλη, της ε, τις ότι χρειάζεται μια αλλαγή, μια εξέλιξη και όχι μια επανάσταση. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Η αρχή που θα κάνουμε είναι να δούμε τι δεν πήγε καλά και να δούμε σε διάφορους επιμέρους τομείς πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να πλουστεύσουμε τα πράγματα. Θα προβούμε σε προτάσεις ε, για την πολιτική συνοχής. Θα ήθελα να μιλήσω για μια σημαντική ιδέα. Χρειαζόμαστε πιο στοχοθετημένη προσέγγιση για το κίνδυνο. Ένα από τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι ότι εκεί που εστιάζουμε τους σπόρους. δεν είναι κατά ανάγκη πιο προβληματική και επικίνδυνη περιοχή. Χρειάζεται μεγαλύτερη αναλογικότητα και διαφοροποίηση, επομένω στο μέλλον. Πολύ σύντομα, να απαντήσω το ερώτημά σας για την αξιολόγηση συμμόρφωσης. Μία από τις ιδέες που εξετάζουμε είναι αν η σημερινή διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Αυτό εξαρτάται από αυτό που είπαν και οι συνάδελφοι, το πόσο θα αλλάξουμε στο μεταξύ το σύστημα. Έχουμε ξεκινήσει μια αξιολόγηση της ε, διαδικασίας αξιολόγησης ε, συμμόρφωσης και το συζητάμε με τα κράτη-μέλη. Η αξιολόγηση που γίνεται ε, στα κράτη-μέλη είναι θετική. Θετικός είναι ο απόϊχος από τα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι η, η διαδικασία συμμόρφωσης είναι καλή διαδικασία. Για τον δημοσιονομικό κανονισμό ε, υπάρχουν πολλές ανησυχίες από την ε, πρόθεση που θεωρούμε μερικοί ότι υπάρχει να ενσωματώσουμε τους κανόνες ε, της γεωργικής πολιτικής. Όχι, δεν ασχολούμαστε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, η ετήσια καθάριση λογαριασμών, καταρχήν. Υπάρχουν δύο πλεονεκτήματα πιθανώς από εκεί. Πρώτον, ότι τώρα, εμείς αλλά και οι δικαιούχοι, πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος της περίοδου προγραμματισμού, δύο με δυόμιση χρόνια μετά το τέλος του, προγραμ... του προγράμματος, για να κλείσουμε τους λογαριασμούς. Αυτό συνολικά μπορεί να είναι 10-12 χρόνια. Και για τους μικρούς δικαιούχους, για τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να περιμένουν όλα αυτά τα χρόνια, είναι μεγάλο διοικητικό άχθος. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μια πιο ενιάυσια διαδικασία, να κλείσουμε τους λογαριασμούς, να πάρουμε τα λεφτά, να τα τσεκάρουμε και να πούμε τελείωσε. Αυτό θα μπορούσε νομίζω να διευκολύνει τη ζωή των πάντων. Δεύτερον, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εμείς λογοδοτούμε προς το Κοινοβούλιο. Έτσι, ετησίως προφανώς. Και θα πρέπει να βρούμε τρόπους με τους οποίους ο τρόπος που η Κομισιόν εξηγεί τι γίνεται στα κράτη-μέλη προς δημοσιονομική αρχή να είναι απλός και να υπάρχει μια βεβαίωση αξιοπιστία σαφής. Ε, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας έχει ένα απλό τρόπο. Υπάρχουν και διάφορα, ε, διάφοροι άλλοι τρόποι και μέθοδοι που λόγω της διαφορετικής φύσης του συστήματος διαφέρουν πάρα πολύ και δεν είναι κατάλληλοι. Αλλά δεν θα πρέπει να τα απορρίψουμε όλα από την αρχή. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης θα ήθελα να πω ότι εκτιμούμε ιδιαιτέρως τις προτάσεις και την αξιολόγηση που κάνατε για την κατάσταση και ε, έτσι έχουμε πλούσια τροφή για σκέψη όλη αυτή την ε, προπαρασκευαστική περίοδο όσο ετοιμάζουμε τη μελλοντική πολιτική συνοχή. Φάνηκε και από τι παρουσιάσει αλλά και από τι αμφιβολίε και του ενδιασμού των συναδέλφων και των μελών της Επιτροπής ότι υπάρχουν διστάμενες απόψεις βέβαια, αλλά πολλά εξαρτώνται και από την εμπειρία που έχει ο καθένας ό,τι αφορά τους τελικού και τους ε, διαφόρους φορείς του συστήματος. Και δεν έχουμε μόνο τις απόψεις ε, των φορέων διαχείρισης ή των ελεκτικών αρχών. Υπάρχουν πολλές απόψεις και πολλές εκτιμήσεις του συστήματος. Και είναι περίπλοκη αυτή η διαδικασία της απλούστευσης. Από μόνη της η διαδικασία αυτή είναι περίπλοκη. Πάντως από αυτά που είπατε κατάλαβα ότι για κάθε λύση υπάρχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και κόστος και όφελος. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη σωστή ε, ισορροπία μεταξύ των θετικών και των αρνητικών σημείων όπως είπα και στην αρχή. Ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή στο σεμινάριο και θα ήθελα μια παράκληση να απευθύνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποια στοιχεία της πολιτικής, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για παράδειγμα, που είναι σημαντική, ή κάποιες διαδικασίες για τις κρατικές ενισχύσεις που χρειάζονται προηγούμενη έγκριση διαφορών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλη αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και δημιουργεί κάποια καθυστέρηση. Οπότε στην προσπάθεια πλούστευσης θα μπορούσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τακτοποιήσει κάπως τα του οίκου της και να επιταχύνει τις εσωτερικές διαδικασίες, να συντομεύσει και κατά ένα έτος μερικές φορές την προθεσμία για την έγκριση κάποιου σχεδίου. Αυτό θα βοηθήσει πολύ τους δικαιούχους. Αυτά ως προς το σεμινάριο. Σας ευχαριστώ θερμά και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και άλλες συνομιλίες στο μέλλον με την εξέταση συγκεκριμένων παραδειγμάτων και τμήματων της, του ρυθμιστικού κανονισμού. Σας ευχαριστώ. And now we, we move... Και θα περάσουμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Ψηφοφορία. Θα ήθελα πρώτα να ελέγξουμε τα μηχανήματα, να δούμε αν λειτουργούν. Παρακαλώ βάλτε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες για μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε για να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. still open. There's still less colleagues who not not everybody voted. Ε, δεν ψήφισαν όλοι. Didn't vote. Δεν ψήφισαν όλοι, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν προβλήματα, κυρία Μπέρτερ, Έχω χάσει την κάρτα μου. Εγώ θα σηκώνω το χέρι στην ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εντάξει, επαληθεύτηκε το σύστημα. Σημείο 4. Έλεγχο από τα κράτη-μέλη τη άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τροπολογία 8. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπέρ, παρόλο που δεν ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. Να ψηφίσουμε μαζί τις πρώτες τέσσερις τροπολογίες 8 με 11. Στο σημείο 4 τη ημερήσιας διάταξης ψηφίζουμε τις πρώτες 4 τροπολογίες. Ποιο είναι υπέρ. 8, 9, 10 και 11. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14, 15 και 16 μαζί ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 1. Τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ε, όλες ε, μέχρι το τέλος από κοινού 2 έως 7 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται και με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση άρχεται η ψηφοφορία τέλος 40 ψήφισαν υπέρ ή μάλλον 41 υπέρ μία ψήφος κατά Συγχαρητήρια στο συντάκτη. Α, εγώ ήμουνα η συντάκτηρα της γνωμοδότησης. Αυτό συγχαρητήρια. Πιο δύσκολη ψηφοφορία ε, αφορά το σημείο 5, την ανάπτυξη δυναμικού δημιουργία θέσεων εργασία στο πλαίσιο μια νέα βιώσιμη οικονομία. Αρκετά περίπλοκη και θα είναι και χρονοβόρα αυτή η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα τη τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Ψηφίστε παρακαλώ. Ποιο είναι υπέρ τη συμβαστική τροπολογία 2. Παρακαλώ και πάλι. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ κατά τη συμβαστική τροπολογία 2. Αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Τρία τμήματα. Απαρτίζει τροπολογία. Θα ψηφίσουμε ξεχωριστά. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές και πάλι απορρίφθηκε. Και το τρίτο τμήμα, τροπολογία 14, ποιος είναι υπέρ, 14, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεν προκύπτει με σαφήνεια, ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 14, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 25 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε όχι, εγκρίνεται. Η πέμπτη συμβαστική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτει. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται και αυτή. 30 υπέρ. Όχι 30, έχει καταπέσει. 31, 31 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. με προφορική τροπολογία 31. Θα πρέπει να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, λυπάμαι. Με προφορική τροπολογία, καταρχήν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ της 31 με την προφορική τροπολογία. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39. υπέρ. 39. εννέα, υπέρ. Ε, για τη γλωσσική τροπολογία δεν ψηφίζουμε. Είναι 39 με την γλωσσική τροπολογία, αλλά υπάρχει και υπόλοιπο τμήμα. Θα ψηφίσουμε λοιπόν, δεν είναι μόνο γλωσσική η 39. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40. Ποιος είναι υπέρ, όχι λάθος, όχι 40. 41, 41. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. 51. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον έχει εγκριθεί και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. 41 ψήφι υπέρ, 2 κατά. Μία εποχή. Ωραία. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Συγχαρητήρια στον αρμόδιο. Επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 6. για τη Μαδέρα και τις Αζόρες. Ανταλλαγή απόψεων. και στο τέλος της συζήτησης θα αναγγείλω και την προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Την περασμένη φορά είπαμε ότι χρειάζεται νέα διαβούλευση για τις αποφάσεις που λάβαμε μετά τη θέση ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας και την ανάγκη εισαγωγή νέων ε, άρθρων για τις ε, εκτελεστικές, ε, για τις αρμοδιότητες μετά από εξουδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζαμε, να εγκρίνουμε χωρίς ε, τροπολογίες την πρόταση αυτή, αλλά για να μην δημιουργήσουμε προηγούμενο, προτείναμε να καταθέσουμε κάποιες τροπολογίες, γι' αυτό και ισχύει αυτή η διαδικασία. Θέλουμε και στο μέλλον, αλλά και σήμερα, να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις μελλοντικές ε, τροπολογίες ε, από νομοθετικές ε, δράσεις του Συμβουλίου μετά από ειδική νομοθετική διαδικασία και θέλουμε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία για να υποβάλουμε αυτή την απέτησή μας προς το Συμβούλιο και στο μέλλον να προηγούνται διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τέτοια περίπτωση ο κύριος Τεϊσέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά για την επιμέλεια και την προσήλωσή σας στο θέμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τις περιφέρειες της Μαδέρας και των Αζωρών και υπήρξαν προβλήματα στην νομοθετική διαδικασία, ιδιαίτερα μετά τη θέση και τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα ήθελα να εκφράσω ένα παράπονο και μια δυσφορία για την απόρριψη των προτάσεών μα από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μερικέ από αυτέ κατέθεσα εγώ ο ίδιο και ζήτησα να προσθεθούν στο παράρτημα τη πρόταση κάποια νέα προϊόντα που υπήρχαν στον προηγούμενο κανονισμό του 2008 και που στόχο είχαν να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα των, της Μαδέρας και των αγορών ιδιαίτερα για σημαντικούς οικονομικούς τομείς. Προτείναμε επιμήκυση του καταλόγου με κάποια βιομηχανικά προϊόντα και κάποιες πρώτες ύλες. Δυστυχώς όμως απορρίθηκαν οι προπολογίες που υποβάλαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να εκφράσω λοιπόν ε, το παράπονό μου και τη δυσφορία μου γιατί έχω την αίσθηση ότι και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξαν μια ασυνέπεια για να μην τη χαρακτηρίσω σχιζοφρενική συμπεριφορά. Γιατί τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε κάποιες ε, εκδηλώσεις και με τη χορηγία και του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα Κανάρια νησιά, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε ένα φόρουμ στα Κανάρια νησιά που μίλησε για την ανανεωμένη, ενισχυμένη στρατηγική για τι υπεραπόμακρε περιοχέ, Αυτά στη θεωρία, αλλά στην πράξη όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν αυτή την ενισχυμένη υποτίθεται στρατηγική και τι υπεραπόμακρε περιοχέ, τι βλέπουμε, απόρριψη των προτάσεων και αποφυγή υλοποίησης αυτών των σχεδίων. Άλλωστε, ελάχιστο θα ήταν το κόστος ε, συμπερίληψης και των νέων προϊόντων. Και η προθεσμία είναι και δεκαετής. Λυπούμε, λυπούμε ειλικρινά και θα ήθελα να εκφράσω το βαθύτερο παράπονο μου, τη δυσφορία μου έως και το θυμό μου για τη στάση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το θέμα αυτό. Ελπίζω πάντως ότι θα αυτό το θέμα σήμερα, ώστε να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό, γιατί πρόκειται για τροπολογίες ε, που ευνοούν και τις δύο υπεραπόμακρες περιοχές, και τη Μαδέρα και τις αζόρε. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει να πάρει το λόγο. Έχουμε μια πολύ σύντομη χρονική περίοδο για τις απολογίες μέχρι τις 28 Ιουνίου και θα ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση αρχές Ιουλίου ούτως ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ και για τη ΣΕΡΑ και για τη δική σας εμπλοκή. Μπορούμε να πάμε τώρα στο σημείο 7. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει μια ομάδα εργασίας και οι πολιτικοί μας σύμβουλοι δούλεψαν πολύ εντατικά τις τελευταίες μέρες και σήμερα ακόμα. Ξεκινήσαμε σε επίπεδο συντονιστών την προσπάθεια να ολοκληρώσουμε το έγγραφο θέσης και μετά από αυτή την συνεδρίαση θα αναθεωρήσουμε το σχέδιο του κειμένου με σκοπό να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν, ούτω ώστε να το έχουμε έτοιμο ε, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Περιφερειακής Ανάπτυξης προς επικύρωση. Αυτά και ελπίζω οι συντονιστές αμέσως μετά από τη σημερινή συνεδρίαση να καθίσουν εδώ για να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Αν δεν υπάρχουν σχόλια. Κύριε Αγγουράκη. Κύριε Αγκουράκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο και θέλω απλώ να κάνω μια ε, τοποθέτηση, μια δήλωση. Ε, παρακολούθησα τη συνεδρίαση των ε, συντονιστών ε, σήμερα το μεσημέρι. Και πράγματι πρέπει να αναγνωρίσω ότι γίνεται μια σημαντική δουλειά, σοβαρή δουλειά από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Εμείς ως Γκουε δεν συμμετέχουμε σε αυτή την ομάδα, όπως γνωρίζετε, και δυστυχώς δεν μπορούμε να συμβάλλουμε στην επεξεργασία αυτού του κειμένου για τους εξής τρεις βασικούς λόγους. Πρώτα απ' όλα το κείμενο αυτό κινείται στη στρατηγική της Λισαβόνας και τη στρατηγική του 2020 που η ομάδα μας δεν συμφωνεί και την έχει καταψηφίσει όπως γνωρίζετε